Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Καλή σας μέρα πρώτα απ' όλα. Αν δεν υπάρχει λοιπόν καμία παρατήρηση σχετικά με την ημερήσια διάταξη, θεωρούμε ότι εγκρίνεται αυτή η ημερήσια διάταξη σε μια αντιπροσωπεία από την Bundeswehr. Ε, στελεχών ε, ευχόμαστε το καλώς ε, ήλθαν και για το χρονοδιάγραμμα στις 28 Σεπτεμβρίου Μαζί με την ΕΦΕΤ θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα έχει να κάνει με το σημαντικό θέμα της συνέχισης αυτής της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας σε κοινό κοινοβουλευτικό πλαίσιο. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά και διάφορα αντιφατικά και γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να είστε παρόντες αν μπορείτε βέβαια στη συνάντηση αυτή και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις που έδειξαν ότι συμφωνούσαμε σχετικά με τις προτάσεις του Άντρου του συναδέλφου και απέναντι δε και στους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να επαναλάβουμε και σημαντικό είναι αυτό, τις θέσεις μας επί του θέματος. Σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με ένα θέμα που ήταν επίκαιρο του τελευταίους μήνες αλλά μας απασχολεί ακόμη με μακρύτερο χρονικό διάστημα και δυστυχώς δεν μπορούμε να το εξετάσουμε για λόγους οργανωτικούς νωρίτερα την ασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ και ε, με την κρίση των ομήρων και τον τραγικό θάνατο ενός ε, Γαλλομήρου και ευτυχώς δύο Ισπανοί ομήροι απελευθερώθηκαν, έχουμε και άλλους όμως εκεί και βλέπουμε ότι και πάλι είχαμε καινούριε απαγωγές ζωπηρώθηκε ε, μπορούμε να πούμε το φαινόμενο αυτό και όλα αυτά είναι γενικά φαινόμενα όπως το είπε ο πρόεδρος του Μαλή την προηγούμενη εβδομάδα στο που νομίζω ότι όλοι μας την προσέξαμε και... νομίζω ότι είναι στα πλαίσια της κοινή λογικής ε, στα πλαίσια αυτών των μέσων που, προσφέρονται από τη συνθήκη της Σαββόνας ε, και ευτυχώς ε, ε, χαιρόμαστε που είμαστε χαίροι γιατί έχουμε τα εργαλεία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερα γάμα μέσων ε, που μπορούμε να προσφέρουμε σαν βοήθεια απέναντι στην περιοχή του Σεχέλ και στα πλαίσια μιας κοινή στρατηγικής, όπως μας υπενθυμήθηκε δε, όλοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε προκλήσεις και ακόμα τα θέματα της ασφάλειας άμυνας δεν έχει να κάνει μόνο με τους ομήρους αλλά βλέπουμε ότι κυκλοφορούν ναρκωτικά όσο ποτέ στο παρελθόν ανθρώπων, ε, όπλων και τρομοκρατικές καθαρά δραστηριότητες. Εδώ και αρκετά χρόνια οι οργανώσεις ε, οι τοπικές, ε, συμφωνώντας με την Αλκάιντα κλπ. Έχουμε οργανώσεις που συνδέονται, συνεργάζονται άμεσα με την Αλκάιντα και αυτό αποτελεί βέβαια μια απειλή άμεση για τις χώρες της περιοχής αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη της ακριβώς να κατανοήσουν όλοι τον κίνδυνο που προκύπτει από όλα αυτά. Έχουμε τρεις ε, προκεκλημένους που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή και τα προβλήματά της, τον Ζίλντερ Κερκόφ, συντονιστή αντιδημοκρατικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πολύ συχνά είναι παρόν στην περιοχή αυτή. Λόπες Μπλάνκο στην Κοινική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε, και παρόν αρκετά συχνά και εκεί. Η κυρία Σεσίλια Ρόστρομ Ρόιν, πεσταμένη του κλάδου πρόληψη τρομοκρατία του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών και για τον έλεγχο των ναρκωτικών ε, θα μπορούσε να ξεκινήσει τη συζήτηση ο κύριος Ντεκερκόφ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία σας αυτή, την οργάνωση αυτής της συζήτησης και για την προσκλησή σας επίσης. Πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα, σημαντικό, κάτι το επίγον για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και της περιοχής του Σαχέλ επίσης, τα κράτη δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα ξεκινώντας να πω στα γρήγορα ποιες είναι οι απειλές, ποιες είναι οι προκλήσεις, όπως επίσης και οι γεωπολιτικές και θεσμικές προκλήσεις ακριβώς που αντιμετωπίζουν οι χώρες στην περιοχή να σας πω ποιες είναι οι προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσφέρει σε αυτές τις απειλές και σε αυτές τις προκλήσεις απαντήσεις. Να αναφέρω μερικά θέματα και το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, οι εκπρόσωποι και ο Επίτροπος επί της Ανάπτυξης τις επόμενες εβδομάδες πώς θα μπορούσαν να τα εξετάσουν για την αυτό για να έχουμε μια συγκεκριμένη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυσκολίες, απειλές, προκλήσεις. Για τις απειλές το είπατε, συντομία. Η περιοχή του Σαχέλ ε, αντιμετωπίζει αυτό το εκρηκτικό μείγμα απειλών με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν, όχι μόνο τη βοκαίνη αλλά και το χασίς και βλέπουμε τις διάφορες οργανώσεις εκεί, τις νοτιοαφρικανικές κυρίως, αλλά και κολομβιανές να χρησιμοποιούν τη Δυτική Αφρική, αλλά έχουμε και διαδρόμους, είδαμε και ε, στο Μαλί που προσγειώθηκε με δυσκολία ένα ε, αεροπλάνο και και επίσης όπλα και σιγαρέτα. Ε, λοιπόν, η Ισπανία στη Μαυριτανία έχει καταβάλει πολλές προσπαθήσεις και τη τρομοκρατία ακριβώ το είπατε, το ε, της Αλγερίας ε, συνεργάστηκε με την Αλκαϊντά και την Κατυπιόντα στην περιοχή του Μαλή με διάφορες δραστηριότητες κυρίως στη Μαυριτανία και στην Νίγηρα κάπως και με τις περιοχές κυρίως της Μαυριτανίας. Θα επανέλθω δε για να δούμε πώς έλαβε ριζοσπαστικό χαρακτήρα αυτή η δραστηριότητα στη Μαυριτανία και πώς ε, έχουμε παγώγης ε, σε 1,5 χρόνο 11 Ευρωπαίων. Ο Μισελ Ζερμανό βλέπουμε ότι βρήκε το θάνατο και ο Βιντάιερ επίσης λίγο νωρίτερα, ε, Βρετανός και με λίτρα ζητούν και μέχρι και 40-50 εκατομμύρια δολάρια λένε οι αλλιερινές ε, αρμόδιες υπηρεσίες και ήδη τα δύο εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή αυτή είναι τρομερό ποσό και μπορούν να αγοράσουν τη σιωπή των τοπικών πληθυσμών, να αγοράσουν ε, τζιπ, ε, ε, όπλα κλπ. Λοιπόν, έρευνες και επαφές με το βρατούν και βλέπουμε την ένταση που υπάρχει ανάμεσα σε χριστιανούς και σε μουσουλμανούς, την σέκτα του Αχάμ ιδιαίτερα ζησπαστικής τάση και επίση ε, για την εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, πόσο συνδέονται αυτό όλα αυτά, απασχολεί τι ε, μυστικέ υπηρεσίε και της Γαλλία και της Ισπανία και ε, βέβαια όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Έχουμε διάφορου πυρήνε οργανωτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρουμε, και αυτό μας απασχολεί στις υπηρεσίες πληροφοριών, αυτοί οι πυρήνες που οργανωτικά με χρήματα και ε, διάφορες ταυτότητες και λοιπά διαβατήρια εφοδιάζει. Το 97 στη ΓΕΑ στο Παρίσι, βλέπουμε τι έγινε, ότι είχαμε επιθέσεις στην Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις απειλές και οι περίπλοκες είναι οι σχέσεις όλων αυτών και με τον Λόπες Μπλάνκο, τον συνάδελφο, πήγαμε σε αυτές τις χώρες και δύσκολο, πολύ δύσκολο είναι ανάμεσα στην ε, Ισλαμική οργάνωση και τον, το οργανωμένο έγκλημα και τον τόπιο πληθυσμό. Δεν ξέρουμε ποιος είναι με ποιον και τι σχέση έχει ποιος με ποιον. Κάτι ακόμα που μας απασχολεί περισσότερο είναι ότι έχουμε δύο περιοχές κρίσης της ε, ΧΕΛ και έχουμε και στη Δυτική Αφρική την περιοχή με πωλήση κοκαίνες, κυκλοφορία κοκαίνες και ε, όπως στη Γουινέα Μπισάου την απειλεί ιδιαίτερα το φαινόμενο αυτό, καταστροφικά τα αποτελέσματα επιπτώσεις. Και βλέπουμε διάφορες προσπάθειες με διάφορους που τα υποστηρίζουν αυτά και από το εξωτερικό. Ένα ε, οι μαλιχίτες, οι σούφοι, πώς θα αλλάξουν και θα γίνουν περισσότερο ριζοσπαστικοί, οι ακραίοι. Και βλέπουμε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν εκατομμύρια χιλιόμετρα ερήμου και έτσι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια ασφαλιακή. Υπάρχει φτώχεια, ξηρασία, ε, κρίση για τα τρόφιμα, πείνα σε πολύ κόσμο στον Νίγηρα και επίσης ένα μέρος στη Μαυριτανία, στο Μαλίκη και Κάτι δε εκεί να προσθέσουμε. Επικρατεί έτσι ανάμεσα στους Άρεγκ και ένας εκνευρισμός, γιατί στην Ήρια η Λιβύη και το Μαλί από την άλλη μεριά υπάρχουν προσπάθειες από αυτούς για επαναστατικά κινήματα. Ε, αυτά όμως δεν ήταν καλοργανωμένα και το ΆΡΕΓ είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με όλα αυτά. Σε αναστάτωση βρίσκονται και υπάρχει μια ένταση και ανάμεσα στις διάφορες φυλές, ανάμεσα στο ΆΡΕΓ, τους Σανγκάι, τους Άραβες, του Αρεγόλους όλους ε, και υπάρχει και διαχείρισης, διακυβέρνηση σε ένα σοβαρό πρόβλημα και είχαμε και στον Ήγερα, τώρα τελευταία μόνο το επισκεφθήκαμε γιατί υπήρξαν προσπάθειες και και κλπ. Και τώρα τελευταία ε, είχαμε περισσότερη ασφαλεία στην περιοχή. Αυτές οι απειλές και αυτές οι προκλήσεις κάνουν, ε, δημιουργούν μια περιοχή περισσότερο εύθραυστη, κλιμακώνεται όλο αυτό γιατί ε, με την τρομοκρατία ε, δεν έχει πια τουρισμό. Ξέρουμε όμως ότι ο πληθυσμός θα μπορούσε να ευνοηθεί από τις τουρίστες, κρίση στο κράτος. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κλιμάκωση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αυτό δίπλα στην Ευρώπη και τις 25 Αυγούστου ο πρόεδρος Σαρκοζή στη διάσκεψη των πρέσβεων είπε ότι τα στενά του Γιβραλτά αναπέχουν 12 χιλιόμετρα μόνο, κοντά κοντά δηλαδή. Άρα λοιπόν και μετά από αυτά δυσκολίες γεωπολιτικές. Τι γίνεται εκεί, το πλαίσιο το περιφερειακό για να ασχοληθεί κανεί με αυτό έχει χαρακτηριστεί με μια μεταβλητή γεωμετρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί δεν συμμετέχει το Μαρόκο. Η ΣΥΝΤΕΟ δεν συμμετέχει εκεί η Μαυριτανία. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από όλου στην περιοχή. Άρα λοιπόν και υπάρχουν και συνδυασμοί από την άλλη μεριά, η Λιβύη, η Αλγερία με χειρισμούς διάφορους ε, και έχουμε και τη Δυτική Σαχάρα. Το θέμα εκεί δεν έχει λυθεί και λοιπόν μπερδεύουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, Ακριβώ είπατε κι εσείς ότι είναι κατεπήγον ο χαρακτήρας. Χρειάζεται μια ανάλυση και μια προσπάθεια της Ευρώπης για να λυθούν αυτά τα πράγματα και από την Ευρώπη πριν να είναι πολύ αργά. Για να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα ένα ενάμιση χρόνο από τότε η Γενική Διευθυνσία Ανάπτυξη Λόπες Μπλάνκο ε, και εγώ ίδιος ε, με την Προεδρία της Σουηδική και την Ισπανική τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, να προσδιορίσουμε μια στρατηγική ασφάλειας και ανάπτυξης. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο ιδιαίτερα να επιμείνω. Ήταν από αυτά που με ανησυχούσαν στο ξεκίνημα αυτής της πορείας τι γίνεται, χωρίς κανείς να λέει τι πιστεύει, να δίνει σημασία στο τι πιστεύει ο καθένας, αλλά η δική μας η δεν είναι ε, μόνο ασφάλεια, αλλά κάτι το περισσότερο σφαιρικό. Αλλά τι γίνεται, νομικά και γεωπολιτικά τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, νομικά, εσείς ε, ε, μιλήσατε κατά της Επιτροπής, γιατί στην Ασία με κονδύλια από την ανάπτυξη εκεί αφιέρωσαν εκείνη αυτά τα χρήματα και γι' αυτό δυσαρεστηθήκατε με την Επιτροπή. Θα πρέπει κανείς όμως να προσέχει για να μπορέσει να πετύχει και στο στόχο το 0,7% του ΑΕΠ για την βοήθεια στην ανάπτυξη και σίγουρα υπάρχουν και συγκεκριμένοι υπολογισμοί στον ΩΣΑ για να δούμε τι γίνεται, τι μπορεί να έχει κανεί την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Ο στόχο πάνω απ' όλα είναι όμω ε, η μάχη κατά τη φτώχεια και όχι η μάχη κατά του εγκλήματο. Τι γίνεται, χρειάζεται όμω ε, κάτι το γενικό σφαιρικό. Χωρί ασφάλεια δεν έχουμε ανάπτυξη. Αν πάτε στο βορρά του Μαλή δεν υπάρχει κανεί που να συνεργάζεται εκεί γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί να τον απαγάγουν. Χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει ασφάλεια και μακροπρόθεσμα. Στην Κιντάλ, στην περιοχή αυτή οι κάτοικοι επαγγελματικά τι μπορούν να κάνουν Εντάξει, η λαχμή από τη στιγμή που έχει χρήματα τους δίνει δυνατότητες άλλων δραστηριοτήτων και πρέπει να, πάμε, να είμαστε εκεί, να δούμε τις δυνατότητες και να κινητοποιήσουμε οποιαδήποτε μέσα, εργαλεία για σταθερότητα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης κάνει μια εκτίμηση, με ένα προγραμματισμό αυτό του 15ου και θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να δούμε πού μπορούν να πάνε για να βελτιώσουμε την ανάπτυξη και την ασφάλεια μαζί. Δεν επιθέτω σε λεπτομέρειε των προγραμμάτων τα οποία πραγματοποιούνται, σχεδιάζονται. Με ένα παρα... μερικά παραδείγματα όμως. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες για την ασφαλεία, τη δικαιοσύνη, τον έλεγχο στα σύνορα. Αυτό και στο Μαλί και στη Μαυριτανία δεν είδαμε ακόμα κάτι συγκεκριμένο για τον Ήγηρε, γιατί ε, είπαμε ότι μετά από, την... Ε, μετά από την αλλαγή προς δημοκρατικό καθεστώς να δούμε τη βοήθεια προς την ανάπτυξη και στον Μπαμακό να ε, έχουμε μια αντιπροσωπεία, ασχολούνται οι Γάλλοι εκεί μαζί με τη δικαιοσύνη και την αστυνομία για να βοηθήσουν εκεί στην εκπαίδευση οργάνων για την ασφάλεια και στη Μαλή και στη Μαυριτανία με βάση στοιχείων, με καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε όλους που συνεργάζονται και συμμετέχουν. Ένα workshop για ειδικευμένοι κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της δημοκρατίας, όπως ε, το πρότυπο στη Μαδρίτη, είτε ο Πόλος Δημοκρατικό στο Παρίσι, με ειδικό προσωπικό εκπαιδευμένο και με κατάλληλη δικαστική υποστήριξη. Και επίση εργαστήκαμε με γαλλική προτεραιότητα για τα σημεία συνόρων, κυρίως το πέραν συνόρων στη Μαυριτανία. Και κάτι ακόμα που έχει σημασία, θα επανέλθω σε λίγο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Μαλή για να αναπτυχθεί στο βόρειο Μαλή με το σχέδιο το κύριο που αναπτύσσεται εκεί οι στατικές βάσεις στο Βόρειο Μαλί να λειτουργήσουν με βάσεις κρατικές που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με την υγεία και διοικητικά, διοικητικές δραστηριότητες. Τώρα να δούμε. Ένας ε, κάτοικος του Κιντάλ ε, πιο εύκολο να πάει στην Αλγερία, στο Αλγέρι παρά στην ίδια την πρωτεύουσά του. Ε, αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάτι το σίγουρο εκεί. Επισχέδια για τους νέους, εκπαίδευση για αυτούς, για δυνατότητες επαγγελματικές, είπα ότι είναι κατεπήγον αυτό. Και επίσης την όλη διαχείριση διακυβέρνηση, μια αποκέντρωση, μήνυμα που μας δόθηκε όταν πήγαμε στον Ήγηρα, ε, να λαμβάνονται αποφάσεις όσο γίνεται περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα επιτόπου, με διαφάνεια στην εξαγωγή των ε, ορεικτών ε, καταλαβαίνετε το πρόβλημα που υπάρχει εκεί και καλύτερος διάλογος ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες. Και επίσης να δούμε τα υπόλοιπα όλα αυτά που θα πάνε στις 5 Οκτωβρίου στην Επιτροπή για την Άμυνα και την Ασφάλεια και κανονικά, αλλά δεν έχει ληφθεί ε, απόφαση για να ληφθεί τελική απόφαση αργότερα κάπως ίσως 25 Οκτωβρίου από τους Υπουργούς Αρμόδιους. Έχουμε τώρα την τεχνική πρόοδο και εκεί αρκετή έχει επιτευχθεί. Ήρθε η ώρα για να προχωρήσουμε σε μια κινητοποίηση πολιτική εκεί, πέρα από την καθαρή πολιτική, ε, τεχνική αρρωγή. Να δούμε πολιτικά τα πράγματα, γιατί διαφορετικά ίσως θα είχαμε μια κρίση ασφάλειας περιφερειακή και θα ήθελα να αναφέρω τρία θέματα, τρία συν δύο θέματα και δεν φαίνονται καθαρά οι απαντήσεις ποιες μπορεί να είναι και θα πρέπει κανείς να τις αναλύσει λεπτομεριακά. Κάτι που με απασχολεί εμένα πρώτα απ' όλα είναι να δούμε πώς ε, στο Βόρειο μαλή θα επικρατήσει και πάλι κρατικός έλεγχος ε, γιατί στις τρεις χώρες ε, που επισκεφτήκαμε είδαμε ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα από το Μαλή να ξεκινήσουμε. Βέβαια, ε, βλέπουμε τι έχει γίνει στο Βόρειο Μαλή. Ε, πρέπει να ξεκινήσουμε από μια τεχνική ανάπτυξη, αλλά και κάτι περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα, το πρώτο ερώτημα. Και η περιφερειακή συνεργασία, πώς να ενθαρρυνθεί. Για περιφερειακή απειλή χρειάζεται περιφερειακή απάντηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα όμως, γιατί δεν υπάρχει ανάμεσα στις ντόπιες κοινότητες μια εμπιστοσύνη. Και ο πρόεδρος είπε ότι ε, πάνω από δύο χρόνια υπάρχει μια διάθεση στον Παμακό να υπάρξει μια σύσκεψη για την περιφερειακή πολιτική. Τι γίνεται όμως με την Αρλεσιανή, που, την όπερα που όλο την περιμένει κανείς όλο το έργο και ποτέ δεν φτάνει μέχρι το τέλος. Λοιπόν, επίσης ε, δεν υπάρχουν δυνατότητες τόσες. Ε, πριν να πούμε ναι, μια διάταξη περιφερειακή και να υπάρξει ένας πυρήνας ασφάλειας ε, στη Σαχέλ που θα υπάρχει για τους αστυνομικούς των τριών κρατών μια κατάρτιση, μια εκπαίδευση. Τι γίνεται, δεν μπορεί το κάθε ένα κράτος για φορτικά να συμμετάσχουν μαζί, δεν ξέρουμε αν είναι η καταλληλότερη λύση. Τι γίνεται, να μπερδευτούν όλοι αυτοί ε, ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να γίνουν σε περιφερειακό επίπεδο ή σε κάθε κράτο. Και η Αλγερία ανέβη μια πρωτοβουλία του 7, υπουργό εξωτερικών, Αλγερία, Βουλκίνα Φάζα, Μαλή, Μαυριτανία, Μαυριτανία-Νίγηρα ε, τη 16 Μαρτίου που μα πέρασε, 4, Απριλίου η επικεφαλή των υπηρεσιών ε, πληροφοριών και στο το γενικό επιταλείο, ας το πούμε έτσι, με τη συμμετοχή αυτών των κρατών συνεδρίασε. Είναι μια αρχή μόνο αυτό. Αν δεν επικρατεί εμπιστοσύνη, δεν θα ενημερώνουν στον άλλο κατάλληλα. Για να δούμε τώρα άλλο θέμα. Τι θα μπορεί να αντικοποιήσει με τα κράτη αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση το διάλογο. Θα πρέπει να ξεκινήσει ένα άμεσο απευθεία διάλογο για την ε, άμυνα, την ανάπτυξη Μαλή, Νιγήρα, Μαυριτανία και αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια τη Αφρικανική Ένωση ε, και τα κράτη Μαγκρέμπ να συμμετάσχουν. Ε, δύσκολο είναι να απαντήσει κανεί Δύο τελευταία θέματα και ολοκληρώνω. Το πρώτο δεν είναι ερώτημα, δεν ε, μια ανάγκη είναι πρέπει διμερός να βελτιώσουμε την οργάνωσή μα Και πέντε δέκα κράτη συμμετέχουν στι προσπάθειε μέρου αυτού του κόσμου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα για τα μέτρα που αποφασίζουμε και με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ο Καναδά που θα αφιερώσει αρκετά χρήματα και επίση οι ΗΠΑ, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στι ΗΠΑ και με του ομολογούς μου ε, συναντήθηκα και τους απασχολεί ιδιαίτερα τους Αμερικανούς το θέμα του Σαχέλ. Ένα δεύτερο σημείο και αυτό είναι σημαντικό αυτό που είπατε για τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρξει μια ομοφωνία με συγκεκριμένη σφαιρική δράση. Ο κύριος Ορτοφέη και ο κ. ο Υπουργός Εταιρικών της ε, Εξωτερικών ε, Υπουργοί να δούμε πώς θα πετύχουμε μια συμφωνία για τη διεθνή κυκλοφορία μάλλον ε, επιτέθη μια συμφωνία τον Ιούνιο για ε, στο Γκάνα, στο Ντακά να δούμε με, με τη Λισαβόνα μαζί και με την ε, Τουλόν να έχουμε μια συνεργασία κατά των ναρκωτικών και με τη συμμετοχή του πρώην τρίτου πυλώνα για να μπορέσουμε, επειδή υπάρχουν δύο περιοχές, να έχουμε μια προσέγγιση ολοκληρωμένη για την ασφάλεια, για την εσωτερική ασφάλεια, για την άμυνα. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση το Αυτά θα σας πω ξεκινώντας τη συζήτησή μας και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ όλοι ο κύριος Λιμπλάν που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα. Εκτιμώ όλου ιδιαίτερω που βρίσκομαι εδώ με του συναδέρφου, που σίγουρα οι γνώσει του είναι πολύ καλύτερε από τι δικέ μου για το θέμα. Γι' αυτό και δεν έχω να προσθέσω, η αλήθεια είναι πάρα πολλά σε αυτά που είπε ο Ζήλ. Γιατί ειλικρινά πάρα πολύ καλά περιέγραψε τη διάγνωση του θέματος. Στη δικιά μου την παρουσίαση θα υπάρξουν βέβαια κάποιες αποχρώσεις αυτά που είπε ο αλλά μια που 1,5 χρόνο συνεργαζόμαστε μαζί πάνω σε αυτή την υπόθεση, καταλαβαίνετε ότι έχουμε κοινή αντίληψη των πραγμάτων. Θα ξεκινήσω λίγο με την προβληματική. Όπως είπε και εκείνος, τα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι ότι πρόκειται για έναν ωκεανό. Μπορούμε δηλαδή να πάμε από οπουδήποτε, οπουδήποτε αλλού, με χίλιους δυο τρόπους. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη όσον αφορά την κυκλοφορία. Μπορεί να έχουμε οποιοδήποτε είδους κυκλοφορία εκεί. Και είναι ένας ωκεανός με ελάχιστη παρουσία κρατών. Είναι μια περιοχή εκτός δικαίου, και με κράτη το οποίο είναι πολύ αδύναμα και εύθραυστα. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε εύθραυστα σύμφωνα με τον τελευταίο ορισμό του τι είναι εύθραυστο, δεν είναι μαλλί, δεν είναι γουνέα μπισά, παρόλα αυτά, ναι. Έπειτα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιβάλλουν την κυριαρχία τους πέρα από τις πρωτεύουσές τους. Και κυρίως πηγαίνοντας βόρεια, αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Η αδυναμία αυτή, σε έναν κάποιο βαθμό, απορρέει από πολιτικούς διακανονισμούς που είχαμε κατά το παρελθόν. Η μη παρουσία των ανθρώπων του Μαλή στο Μαλή οδήγησε και σε αυτά που έγιναν με του ΑΡΕΚ τη δεκαετία του 90. Το κράτος παρετήθηκε από την παρουσία του εκεί για να αποφύγει τα προβλήματα με το Στουαρέκ. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώς συνοψίζουμε την κατάσταση σήμερα και τι κάνουμε σήμερα, μην δημιουργήσουμε προβλήματα άλλα στο μέλλον. Η περίπτωση του Μαλή είναι πολύ χαρακτηριστική γι' αυτό. Αυτό έγινε στο παρελθόν. Αυτή λοιπόν η αδυναμία, η μη παρουσία των κρατών, τα χαρακτηριστικά της περιοχής, Σαχάρα, Σαχέλ, που δεν ελέγχονται, δεν υπάρχει δυνατότητα, οδήγησε σε ένα πεδίο γόνιμο για την εγκατάσταση της ΑΚΜΗ στο βόρειο Μαλή, της οργάνωσης αυτής, η οποία γεννήθηκε και προέκυψε όχι από εσωτερικά προβλήματα των δύο χωρών που εξετάζουμε εμείς, έρχεται απ' έξω, είναι εξωγενής. Η ΑΚΜΗ είναι μια οργάνωση εξωτερική, εκτός των τρών περιοχών στην περιοχή, που προσπαθεί όμως να ριζωθεί, που προσπαθεί να δημιουργήσει ρίζες εκεί. Είναι κλασική τεχνική γάμη με τοπικό πληθυσμό, αγορές, Αγοράζει ένα πρόβατο από την Αλκαίδα που το πληρώνεις τρεις φορές παραπάνω από ό,τι στην ε, αγορά. τεχνική που κάνει την Αλκάιντα να θέλει να είναι παρούσα στο Μακρέβ. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν είναι μια παρουσία εκεί με, στρατηγική η ειρηνικά να εγκατασταθεί. Υπάρχει εκεί ακμίδο και 20 χρόνια. Και πρόσφατα από το 2005 δεν υπήρξε επίθεση στην τρομοκρατική επίθεση στη Μαυριτανία. Από το 2005. Αλλά η ΑΚΜΗ ήταν ήδη εκεί στη Μαυριτανία πολύ πριν. Άρα λοιπόν η στρατηγική τους είναι παρουσία προκειμένου να ριζωθούν στην περιοχή με επαφές με τον πληθυσμό, κάτι το οποίο βλέπουμε και αλλού εξάλλου. Το πρόβλημα θα είναι Πώς θα κόψουμε αυτή τη σχέση με τον τοπικό πληθυσμό που υπάρχει. Ποιος είναι ο μηχανισμός που μπορούμε να βρούμε ώστε η ακμή, παρόλο που προσπαθεί να έχει τέτοιες σχέσεις με τον τοπικό πληθυσμό, εμείς πώς αυτές τις σχέσεις θα τις κόψουμε. Βέβαια εύκολα λέγεται και πολύ πιο δύσκολα γίνεται. Όπως είπε και ο Ζήλτε Κερκόβερ, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε, η Γενική Γραμματεία δηλαδή του Συμβουλίου, οι συντονιστές, η Επιτροπή, η ΕΣ, η Προεδρία, τα κράτη-μέλη, αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Μια στρατηγική που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και καλά το σκεφτόμαστε, αλλά θα πρέπει πρώτον να καταλήξουμε σε μια κοινή διάγνωση για το πρόβλημα. Να συμφωνήσουμε για τη διάγνωση αυτή. Και δεν φτάνει κιόλα. Είναι αναγκαίο, αλλά δεν φτάνει. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία δράσης. Όπως είπε και ο Ζίλντε Κερκόβε, αναπτύξαμε πρώτα απ' όλα έναν ρόλο επιλογής. Παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο. Λέμε δηλαδή ότι θέλουμε να εξετάσουμε πρώτα τους παράγοντες κινδύνου. Τι παράγοντες κινδύνου υπάρχουν και κατά πόσο είναι περιφερειακής φύσης ή όχι. θέλαμε να αποφασίσουμε κατά πόσο πρόκειται για προβλήματα στην περιοχή, για εθνικά ή όχι. Δηλαδή το Αρέγκα στο Μαλί και στη Μαυριτανία συνδέονται, έχουν κοινά προβλήματα. Τι είναι γκάρσιο δηλαδή στην περιοχή. Αλλιώς δεν χρειάζεται να μιλάμε για περιφερειακή στρατηγική, θα εξετάσουμε τα προβλήματα τη κάθε χώρα χωριστά. Όχι όμω. θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν εγκάρσιοι παράγοντες. Γι' αυτό και η Επιτροπή δέχτηκε την πρόταση να, κάνει, να έχει μια αποστολή επιτόπου ερευνητική για να δει τι μας λένε οι εταίροι μας για τα προβλήματα εκεί. Και ήταν ξεκάθαρο το ότι βγήκε. Αυτό που όλοι μας είπαν, με τέτοια λόγια περίπου, είναι ότι δεν είναι πρόβλημα που μπορεί μεμονωμένα να λυθεί, ότι είναι περιφερειακό. Μας το είπαν όλοι, σε όλα τα επίπεδα. Ε, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί, επιθεωρητές αστυνομίας, κοινωνία των πολιτών. Ήταν το leitmotiv. Αυτό ακούγαμε συνέχεια. Δεν είναι κάτι που μπορεί μία χώρα από μόνη της να αντιμετωπίσει. Άρα ήταν αναγκαία, μας είπαν, να έχουμε μία περιφερειακή προσέγγιση. Βέβαια, δεν είναι σίγουρο ότι όλοι θέλουν την ίδια περιφερειακή προσέγγιση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί ακόμα και αν έχουμε τέσσερα μεγάλα προβλήματα που είναι η παρουσία της ακμή, τα εγκληματικά δίκτυα που υποφελούνται, οι άνθρωποι που αντιδρούν, η Τουαρέκ ή τα προβλήματα διακυβέρνησης, ο Ισλαμισμός ο ριζοσπαστικός που προχωράει. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα και το ερώτημα που τίθεται, πώς η μία ή άλλη χώρα βλέπει αυτές τις προτεραιότητες, πώς τις ιεραρχεί αυτές τις ε, απειλές. αλλού η ακμή είναι πολύ ψηλά ως προτεραιότητα, αλλού στο Μαλί α πούμε δεν επιτίθεται και δεν είναι. Για πολύ η κυβέρνηση του Μαλί δυσκολευόταν να μπει στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Για να το πω έτσι. Έπειτα ο ριζοσπαστικός Ισλαμισμός το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Είναι κάτι που αγνοήθηκε, υποτιμήθηκε για πολύ καιρό από όλους. Το Ισλάμ ε, είναι ενωμένο, με ανοχή κλπ. κλπ. Και μετά, σιγά σιγά, καταλάβαμε ότι τα τρία τελευταία χρόνια τα ε, ριζοσπαστικά τζαμιά πολλαπλασιάστηκαν επί τρία. Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι υπάρχει μια έκρηξη και στις τρεις χώρες. Όμως εξακολουθεί να ισχύει η άποψη που λέει ότι όχι, είναι ανεκτικό αυτό το Ισλάμ, δεν αποτελεί απειλή και τέτοια. Τώρα βέβαια, ποια ήταν ε, τα συμπεράσματά μας για τις τρεις χώρες, για τη Μαυρετανία πρώτα απ' όλα. Πρέπει να σας πω ότι από τις τρεις ε, χώρες όσον αφορά την αδυναμία, το πόσο έθραυστες είναι. Ακολουθήσαμε το άρθρο 96. Δεν ξέρω κατά πόσο ορισμένοι από σας γνωρίζουν ή δεν το γνωρίζουν. Πάντως το άρθρο 96 βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού είναι μια χώρα ε, που ουσιαστικά κόβεται η συνεργασία είτε λόγω πραξικοπήματος, είτε άλλων στοιχείων που αναφέρεται σε φωνία του Κοτονού. Μαυριτανία πρώτα απ' όλα. Το πρόβλημα διακανονίστηκε και μπορέσαμε να πάμε σε αποστολή εκεί. Ήταν έκτακτη η κατάσταση εκεί για πολύ καιρό και ακόμα η κατάσταση είναι βάση του άρθρου 96, αλλά βρίσκεται σε μια διαδικασία επιστροφής στη δημοκρατία. Γι' αυτό και μπορέσαμε να κάνουμε την αποστολή αυτή με τη συμφωνία βέβαια του Συμβουλίου. Το πλαίσιο δηλαδή βελτιώθηκε κατά πολύ. Είναι όμως ένας δείκτης και αυτός που δείχνει πόσο έθραυστη δημοκρατικά και πολιτικά είναι μια χώρα. Είμαστε λοιπόν στη Μαυρετανία. Πρόκειται για ε, ακραία ένδια, ανισότητες, ε, δυσκολίες στον κοινωνικό τομέα. Οι τρεις ομάδες στον πληθυσμό που είναι οι Άραβες ε, λευκοί, μαύροι, ο πληθυσμός ε, μαύρων εκεί. Δεν βρίσκονται σε συμφωνία για το πώς βλέπουν το nation building. Δεν είναι ξεκάθαρο για αυτούς. Είναι ένα πράγμα που συζητιέται. Φυσικά και υπάρχει μια ελίτ η οποία θέλει μια Μαυριτανία περισσότερο όπως στη Βόρεια Αφρική, Ισλαμική κτλ. Αλλά υπάρχει και μια δημογραφική κατάσταση η οποία πιέζει τη χώρα προς τον νότο. Εδώ δηλαδή κόβεται στα δύο κατά κάποιο τρόπο η χώρα. Γιατί υπάρχουν πραγματικές ανισότητες. Ορισμένοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, είναι μορφωμένοι. Οι θέσεις στο δημόσιο όμως δεν δίνονται πολλές φορές σε αυτούς εξαιτία του ονόματός τους, της πρόλευσής τους. Γι' αυτό, αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω που λέμε ότι είναι έφραυστη η χώρα. Η χώρα βέβαια το γνωρίζει αυτό και προσπαθεί να το λύσει. Δεν είναι κάτι που είναι εκτός της πολιτικής συζήτησης στη Μαυριτανία σήμερα, όχι, είναι κάτι που συζητιέται και που τον αναγνωρίζουν οι ελίτ. Το ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και προσπαθούν να το δουλέψουν και εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Κερχόφε, υπάρχει μεγάλη δυναμία και στο σύστημα ασφάλειας. Και ας υπάρχει στρατηγική για τις ανοπλές δυνάμεις, την αστυνομία κτλ που προσπαθούν με δράσεις να αντιμετωπίσουν ότι δυσκολίες υπάρχουν. Υπήρξαν όμως τρομοκρατικές ε, επιθέσεις. Άρα υπάρχουν ε, πυρήνες, υπάρχουν ε, κέντρα κομμάντος, τα οποία έχουν κάποια βοήθεια προφανώς. Τα κράτη-μέλη μας τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτά από ό,τι πάλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως είναι μια πραγματικότητα αυτή η κατάσταση. Αυτά για τη Μαυριτανία. Μαλή τώρα που είναι ο χώρος όπου είναι και το κέντρο της ΑΚΜΗ. Το κύριο πρόβλημα ήταν η του ΑΡΕΚ και το γεγονός ότι εγκατέλειψε το βόρειο βήμα της χώρας το κράτος. Και αυτό μετά από τη Συμφωνία του 90, το διακανονισμό του 1990. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν ο χώρος αυτός στους του ΑΡΕΚ που θέλανε να τους αφήσουν ε, λίγο αυτονομία και έπεσαν στα χέρια τελικά των διαφόρων τρομοκρατικών δικτύων, της ΑΚΜΗ για παράδειγμα, που δημιούργησε δεσμούς με τον πληθυσμό εκεί. Το πρόβλημα που δεν έχει λυθεί ακόμα ακριβώς είναι οι σχέσεις τώρα των του με το κράτος. Πρόκειται για διαζύγιο που εξακολουθεί. Δεν υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στους Τουαρέκ και την κυβέρνηση, το κράτος του Μαλή. Και αυτό επίσης το εκμεταλλεύονται όποιοι μπορούν. Στο Μαλή μπορούμε να πούμε ότι το κέντρο βαρύτητας είναι κάποιοι τέος μάχημοι οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στην οικονομία οι οποίοι έχουν την τάση, γιατί είναι εύκολο να κερδίσει κανείς χρήματα προστατεύοντας ε, ένα κονβόι με ναρκωτικά ή με κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν συμμετέχουν στην παραοικονομία ή στα εγκληματικά δίκτυα και δημιουργούν επίσης οικονομικά κίνητρα στην παραοικονομία τεράστια. Το είπε και ο Ζήλ πάρα πολύ καλά όταν μιλάμε για ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανασφάλεια, ποιο να στείλουμε. Θα τους απαγάγουν. Πώς να βοηθήσουμε την ανάπτυξη μέσα σε μια τέτοια κατάσταση όταν ελοχεύουν τόσο μεγάλη κίνδυνη. Στη Σομαλία φυσικά είναι πιο σοβαρά τα πράγματα, στην Αφγανιστία, ενώ στο το Αφγανιστάν, το ξέρουμε. Αλλά και στην περιοχή του Σαχέλ είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. δεν στέλνουμε κάποιον εθελοντή να βοηθήσει με χρήματα. Μάλλον, τον βλέπουν σαν ένα σακί ε, φλουριά. Γιατί, γιατί άμα τον απαγάγουν θα μπορέσουν να πάρουν χρήματα. Πιστεύουν. Για τον Ήγηρα. Το ίδιο ισχύει η ανασφάλεια, η ακμή Επίσης υπάρχει και μεγάλη παρανομία. Ε, δεν διακανονίζονται τα προβλήματα με το, το ΑΡΕΓ. Υπάρχουν ε, λοιπόν εκεί οι άνθρωποι που ασχολούνται και με το λαθρεμπόριο, αλλά και πλήττουν την ε, καθημερινή ασφάλεια των πολιτών. Είτε με απαγωγές, είτε κλέβοντας κάποιες αποστολές κλπ. Στο Νίγηρα ο κίνδυνος είναι κυρίως στο βορρά. Πάντως σε σχέση με τις άλλες χώρες, η χώρα αυτή έχει και κάποια σημαντικά στοιχεία. Η αστυνομία και οι δυνάμεις του Νίγηρα είναι σε κάπως καλύτερη θέση από εκείνες του Μαλή και της Μαυριτανίας. Επίσης, ο πληθυσμός συνεργάζεται καλύτερα μαζί τους. Ε, οι διάφοροι τρομοκράτες όταν περνάνε από τη χώρα εκεί πρέπει να το κάνουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλιώς τους πιάνουν, τους βρίσκουν. Στο Μαλή δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ. Δεν τους ε, καταγγέλουν αμέσως. Στον Νίγηρα υπήρξαν περιπτώσεις όπου ο στρατός μπόρεσε και έδρασε τάχιστα γιατί ειδοποιήθηκε. Και από όλες τις χώρες της περιοχής είναι η μόνη που έχει καλές σχέσεις με όλους τους γειτονές της. Με τη Μαυριτανία, με το Μαλί, με την Αλγερία, με τη Λιβύα. Άρα λοιπόν είναι μια χώρα σημαντική για να δημιουργηθεί αυτή η περιφερειακή διάσταση. Τώρα για το πρόβλημα. Πολύ καλά τα είπε ο Υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ των χωρών και με τη διεθνή κοινότητα επίσης. Υπάρχει αδυναμία στα συστήματα ασφάλειας. Ξεκάθαρα. Χρειάζονται ικανότητες που δεν μπορούν να έρθουν μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν με τις δικές τους δυνατότητες και ικανότητες για να βοηθήσουν τις χώρες αυτές. Και το κάνουν ήδη, αλλά πρέπει να το κάνουν ακόμα περισσότερο και πιο συντονισμένα. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι χώρες μέλη έχουν τις δυνατότητες. Και έπειτα είναι πολύ βάλλοντε αυτές οι χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση. Και εδώ είναι και το βασικό ερώτημα του Ζήλ. Πώ να κάνουμε ανάπτυξη σε μια χώρα που επικρατεί η ανασφάλεια. Δεν έχουμε βρει ακόμα λύσει σε αυτό. Πρέπει να δούμε πώς να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα μέσα. Δεν τα έχουμε ακόμα. Επίσης, πρέπει να ασχοληθούμε και με τις διενέξεις που δεν έχουν ακόμα λυθεί. Τα προβλήματα δεν έχουν ακόμα λυθεί όπως είναι το ΑΡΕΚ, όπως είναι τα προβλήματα στη Μαυριτανία. Αν δεν βοηθήσουμε τις χώρες να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα που βρίσκονται σε κρεμότητα, ε, με, αυτά, με αυτές τις πληγές που κάνουν τις χώρες αυτές ε, τόσο ευάλωτες, δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το σύνολο των απειλών. Δεν είναι επειδή έχουμε μια καλή αστυνομία ότι θα λυθεί και το πρόβλημα με του Τουαρέκ. Όχι, χρειάζεται συμφιλίωση. Χρειάζονται δράσει που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Αυτά. Και λυπάμαι αν μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Merci à vous. Ε, Κυρία Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την, για την πρόσκλησή σας. Ε, έχω συντάξει την παρέμβασή μου στα αγγλικά και θα μιλήσω αγγλικά. Θα ευχαριστήσω πρώτα την Επιτροπή σας που προσκαλέσατε την εκπρόσωπο, εμένα δηλαδή, των Ηνωμένων Εθνών, της Μονάδας για, την, ε, για τον μάλλον τον, τον, για του κλάδου για την πρόληψη τρομοκρατίας του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών. Ο στόχος ε, της οργανωσής μας είναι να προσφέρουμε υποστήριξη στις χώρες μέλη για να αντιδράσουν με ε, μέσα κράτους δικαίου στις προκλήσεις που θέτει η τρομοκρατία. Θα σας αναπτύξω τις προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει και στις οποίες ε, χώρες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτές προσφέρουμε τεχνική βοήθεια. Για όσες και όσους εξημών δεν γνωρίζετε το γραφείο μας και τον κλάδο πρόληψης της θρομοκρασίας, ο στόχος μας, όπως είπα, είναι να προσφέρουμε υποστήριξη στις ε, χώρες μέλη μας για να, μπορούν, να μπορέσουν να υπογράψουν και να κυρώσουν τα νομοθετήματα που έχουν, ε, το διεθνούς δικαίου δηλαδή, 168 χώρες έχουν λάβει την υποστήριξή μας από το 2003, όλες οι χώρες του Σαχέλ, επίσης και στην ευρύτερη Δυτική Αφρική και Βόρεια Αφρική. Οι δύο άνδρες που μίλησαν πριν από μένα αναφέρθηκαν στις προκλήσεις για την ασφάλεια και την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Δεν θα ασχοληθώ, θα αναπτύξω λοιπόν περισσότερο το ίδιο το θέμα της ε, απειλής στην ασφάλεια και πώς ορίζεται, αλλά θα τονίσω ότι από την σκοπιά της UNODC η αποτελεσματική απάντηση σε αυτήν την πρόκληση πρέπει να βασίζεται σε αρχές κράτους δικαίου και να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους. Επομένως, μια προσέγγιση δημιουργίας ικανότητας που θα πρέπει να περιλάβει και ε, πρωτοβουλίες στον χώρο της ε, δημόσιας ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της αύξησης της δημόσιας αξιπιστίας των σχετικών θεσμών και την μείωση της διαφθοράς. Το UNODC έχει μια συνολική εντολή η οποία το θέτει σε θέση να μπορεί να βοηθήσει τις χώρες οι οποίες χρειάζονται τη τεχνική υποστήριξη για να ξεπεράσουν τα εμπόδια αυτά. Και σε ό,τι αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας, ε, το, το Terrorism Prevention Branch που εκπρόσωπος είμαι εγώ και που εδρεύει στην Βιέννη αλλά έχει και 25 γραφεία επιτόπου σε διάφορες χώρες. Ε, επίσης έχουμε αξιωματούχους στο Ντακάρ, στο γραφείο μας, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή Σαχέλ. Πάλι από τη σκοπιά του γενόντιση, εμείς εξετάζουμε το θέμα, όπως είπα, σαν μέρος μιας ε, ατζέντα ανάπτυξης και ολοκλήρωσης που είναι συστηματική προσέγγιση στα θέματα αυτά των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη λοιπόν προσεγγίζουν το θέμα με τρόπο παρόμοιο όπως ακούσαμε από τους δύο προηγούμενους ε, ομιλητές και επομένως τα σοβαρά εγκλήματα μεταξύ αυτών και η τρομοκρατία όντως υπονομεύουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η τρομοκρατία ιδιαίτερα αποτρέπει ε, τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν τις επενδύσεις τον τουρισμό και αποτελεί έτσι σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη. Από τη σκοπιά μας εξετάζουμε επίσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και εκεί εκτείνεται η εντολή μας για την ελευθερία διακίνησης, για παράδειγμα την ε, επαγγελματική απασχόληση και τα άλλα δικαιώματα τα οποία όλα υπονομεύει εν τέλει η τρομοκρατία. Στην περιοχή του Σαχέλ ακούσαμε ήδη τις περιγραφές των προκλήσεων στην ασφάλεια που με πολλούς τρόπους δείχνουν κιόλα πόσο σημαντική είναι η εντολή του Ιωνοντισή και η προσέγγιση αυτή. Η διασύνδεση μεταξύ τρομοκρατικών και άλλων εγκληματικών ομάδων στην περιοχή αυτή με λαθρεμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο όπλων που καθιστούν αναγκαίο να υποστηριχθούν οι χώρες αυτές για να μπορέσουν να αντιδράσουν. Από τη σκοπιά αυτή θα ήθελα λοιπόν να ρίξω περισσότερο φως σε τέσσερις επιμέρους προκλήσεις, τις οποίες οι χώρες σε συνεργασία μαζί μας έχουν οριοθετήσει και εκεί χρειάζεται να τις ενισχύσουμε για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Πρώτα, η ανάγκη βασικής επιτόπου εκπαίδευσης, νομικής εκπαίδευσης, για όλους τους αξιωματούχους που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε όλες τις χώρες της ΑΧΕΛ, πολύ λίγοι εισαγγελείς, για παράδειγμα, έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τα πολύ περίπλοκα εγκλήματα που ε, αντιμετωπίζουν εκεί, πραγματικά με πολλές διασυνδέσεις και τρομοκρατικές και ε, με διάφορα εμπόρια κτλ. Δεν υπάρχει εξειδίκευση μέσα στο σύστημα της ποινική δίωξης. Άρα δικαστές και εισαγγελείς διορίζονται για να μπορέσουν να υπηρετήσουν σε οποιοδήποτε δικαστήριο και για οποιοδήποτε θέμα. Ταυτόχρονα υπάρχει σημαντική κίνηση στο, ε, ε, σημαντική κινητικότητα μάλλον ε, ε, στον χώρο τη δικαιοσύνη στην περιοχή αυτή. Άρα οι εισαγγελεί και δικαστέ δεν παραμένουν επί πολύ χρόνο στο ίδιο πόστο. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχυθεί η προσπάθεια των δικαστών και εισαγγελέων. Χρειάζεται επίση να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης όλων όσοι ασχολούνται με θέματα ποινική δικαιοσύνη στην περιοχή αυτή. Αυτά κάνουμε εμείς με, στη συνεργασία με το Μάλι, τον Νίγηρα την Μπουρκίνα Φάσο και, και την τέταρτη χώρα η οποία διέφυγε του Διερμηνέα δυστυχώ. Και προωθούμε λοιπόν συνεργασία με τους θεσμούς σε όλες αυτές τις χώρες ώστε να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες οι ίδιες, οι ίδιοι φορείς και οι θεσμοί επιτόπου και κάνουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ώστε οι εκπαιδευτέ μέσω στους θεσμού αυτούς να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση σε όλους τους δικαστές και εισαγγελεί στην χώρα τους. Πρόκειται για μια προσέγγιση που πολύ θα θέλαμε να δούμε να διαδίδεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, εφόσον βέβαια υπάρξει σχετική χρηματοδότηση. Για την ώρα έχουμε εστιάσει την προσοχή μας σε αυτές τις τέσσερις χώρες που προανέφερα. Θα κάνουμε ένα σε βάθος πρόγραμμα εκπαίδευση των εκπαιδευτών που θα ολοκληρωθεί ήδη πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Δεύτερη πρόκληση, στην οποία αναφέρθηκαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, είναι η πρόκληση και η ανάγκη ενισχυμένης διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας. Αυτό περιέχεται στην εντολή μας και από τη σκοπιά μας, εκεί που δίνουμε ιδιαίτερη σημασία είναι η συνεργασία σε ποινικά θέματα. Η δικαιική συνεργασία δηλαδή, ειδικά σε ποινικά θέματα. Πολύ ξεκάθαρη πρόκληση αυτή στην περιοχή αυτή του κόσμου, όπως εξήγησαν και οι δύο προηγούμενοι, αλλά εκεί επίσης βλέπουμε να γίνεται πρόοδος, αλλά και ξεκάθαρα να υπάρχει η βούληση των ενδιαφερόμενων χωρών να ενισχύσουν την συνεργασία τους. Μετά από εκφρασμένη θέληση των τεσσάρων χωρών, ξεκινήσαμε πρόσφατα μια πλατφόρμα για δικαιική συνεργασία τον Ιούνιο στον Παμάκο. Για δικαιική συνεργασία, δικανική καλύτερα συνεργασία, σε σχέση με την τρομοκρατία, που όμως είναι ενδιαφέρουσα και για την αντιμετώπιση άλλων σοβαρών μορφών εγκλήματος. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν δημιουργήθηκε, όπου οι χώρες αυτές έχουν εκπροσώπους και όπου εμείς παρέχουμε υποστήριξη στις χώρες για να παραγάγουν με τη σειρά τους οδηγούς και εγχειρίδια που να επιτρέψουν τη μετάδοση της γνώσης που είναι απαραίτητη για τα θέματα αυτά. Έχουμε εργαστεί επί χρόνια προσφέροντας υποστήριξη σε διάφορες χώρες για να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία και είναι πολύ θετικές οι εμπειρίες που έχουμε από μια άλλη πλατφόρμα που είχαμε δημιουργήσει των χωρών δηλαδή της Επιτροπής του Ινδικού Ωκεανού. Μέσα σε ένα μόνο έτος κατόρθωσαν οι χώρες αυτές με την υποστήριξή μας να προωθήσουν 30 υποθέσεις ε, αμοιβαία δικαστικής αρρωγής και εν τέλει οι οποίες κατελήξαν σε απελάσεις. Προστιθέμενη αξία των πλατφορμών αυτών είναι ότι αποτελούν βάση για μια κοινή, ένα ε, κοινό μάλλον εντοπισμό περαιτέρω αναγκών ε, χωρίς υποστήριξης. Επίσης, οι χώρες που ξεκίνησαν αυτή την πλατφόρμα Σαχέλ είπαν επίσης ότι θέλουν να παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα αυτή για συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής. Τρίτη πρόκληση, την οποία επιθυμώ να σας επισημάνω, είναι η ανάγκη ειδική υποστήριξης για δημιουργία τεχνογνωσίας σε επιμέρους συγκεκριμένου τομείς που προκύπτει από την διαρκώς ε, μεταλλασσόμενη μορφή της ε, τρομοκρατίας και σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία της και τους στόχους της και τους τρόπους συνεργασίας και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο αναγκάζει τις χώρες να αναπτύσσουν αντίστοιχη τεχνογνωσία σε πολλούς τομείς. Τρεις. Πρώτα, ναυτική τρομοκρατία που είναι όλο και πιο έντονη απειλή στον κόλπο της Γουινέας. Μια περιοχή λοιπόν όπου ο UNODC έχει αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της εντολής του UNODC που έχει σχέση και με την αντιμετώπιση της πειρατείας αλλά και με το ευρύτερο πλαίσιο ναυτικών τρομοκρατικών ενεργειών και αντιμετώπιση τους δηλαδή, προχωρούμε σε στενή συνεργασία και με άλλους φορείς όπως την IMO, τη Διεθνή Ναυτιλιακή Οργάνωση και ε, άλλους παρόμοιους ε, φορείς και θεσμούς. Τον Ιούνιο οργανώσαμε διάσκεψη ε, χωρών της Αφρικής βασιζόμενη στην εμπειρία ότι μεταξύ των χωρών αυτών υπήρχε πολύ περιορισμένη κύρωση, δηλαδή επίπεδο κύρωσης των σχετικών διεθνών εγγράφων. Περιορισμένη επίσης ε, γνώση, επίπεδο γνώσης των θεμάτων, ενώ ταυτόχρονα έχουν πολύ εκτεταμένες ακτογραμμές. Προχωρούμε τώρα στην δεύτερη διάσκεψη για χώρες Δυτικής Αφρικής και Σαχέλ. Μια άλλη πρόκληση αναφέρεται στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επίσης ένας χώρος όπου συνεργαζόμαστε στενά με τις χώρες επιτόπου για να προσφέρουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση. Έγινε για παράδειγμα στον Τακάρ τον Μάρτιο ένα εργαστήρι με ε, χώρες της Δυτικής Αφρικής και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις χώρες αυτές στον τομέα. Κάνουμε, ε, προωθούμε επίσης ε, συνεργασία με ειδικευμένους φορείς, καθώς και με άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έχουμε μια εξαιρετική ε, σχέση εργασίας. Τώρα έρχομαι στην πυρηνική ε, τρομοκρατία, που και εκεί αποτελεί απειλή, και στην περιοχή αυτή αποτελεί απειλή. Υπάρχουν 7 ε, χώρες στην Κεντρική Αφρική που έχουν ουράνιο και που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο τρομοκρατικών επιθέσεων. Τώρα το θέμα είναι εξαιρετικά περίπλοκο, διότι ε, παίζουν ρόλο εκεί διάφορες διεθνή, διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, χρειάζεται δε ε, πάρα πολύ εξειδικευμένη γνώση από αυτούς, αυτών μάλλον που ασχολούνται με το δίκαιο εκεί για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Για να προσφέρουμε τώρα τις εκπαιδεύσεις αυτές, ο Γιάννοντισή στα πλαίσια της πρόληψης χρησιμοποιεί και καινοτόμες μεθόδους, για παράδειγμα επιγραμμικές online μεθόδους ε, εκπαίδευσης με κομπιούτερ κλπ. Και, τις, ε, και για τις χώρες της ζώνης Σαχέλ. Ε, θα προωθήσουμε, θα αρχίσουμε μάλλον τώρα αυτό το μήνα και μια μορφή συνεργασίας στην εκπαίδευση με επιγραμμική όπως είπα που θα συνεχίσει και μετά από την ολοκληρωσή της να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παραμείνουν σε διαρκή επαφή μεταξύ τους. Η τελευταία πρόκληση που θα ήθελα να σας επισημάνω, όπως άλλωστε είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι ότι υπάρχουν ενδεχομένως πολύ στενές διασυνδέσεις μεταξύ τρομοκρατίας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, λαθρεμπόριων ναρκωτικών, τα λαθρεμπόριων ελαφρών όπλων και άλλων δραστηριοτήτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τονιστεί και τα τελευταία δύο χρόνια και από το Περιφερειακό Γραφείο για την Κεντρική και Δυτική Αφρική, του Ντακάρ, του Γιονοντισή και ένα πρόγραμμα εκτεταμένο έχει αναπτυχθεί όπου ο κλάδος πρόληψης ε, του Γιονοντισή παίζει ένα βασικό ρόλο. Από τη δική μας σκοπιά Οργανώσαμε για παράδειγμα πέρσι μια ε, συνάντηση στο Λασπάλμα για τις χώρες του Έκοβας που ζητήσαμε μέσω αυτών δηλαδή από το Γενοντισί να προωθήσει περιφερειακές συνέργειες οι οποίες θα επιτρέψουν ταυτόχρονη πρόοδο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας αλλά και των λοιπόν μορφών του οργανωμένου εγκλήματος με ανάπτυξη κοινών ε, δικαιικών μέσων και Αυτή είναι μια προσέγγιση λοιπόν την οποία προωθεί ο UNODC και όπου ο κλάδος πρόληψης της τρομοκρατίας ως τέτοιος προχωρεί σε μια αποκέντρωση των ικανοτήτων προγραμματισμού και παροχής εκπαίδευσης ώστε να αντιδρά καλύτερα επιτόπου στις ανάγκες που διαπιστώνονται στο ε, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτά τα περιφερειακά προγράμματα υπάρχουν και εθνικά ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία εμπλέκονται. Το πρώτο που αναπτύχθηκε ήταν σε συνεργασία με το Μαλί, με συμφωνία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και η παρόμοια κίνηση σημειώνεται και σε συνεργασία με τις άλλες χώρες. Εν τέλει, όπως είπα προηγουμένως, Έχουμε τις εταιρικέ σχέσεις, συνεργασίες που έχουμε με διαφόρους φορείς για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες διασυνδεόμενες μορφές εγκληματικών ενεργειών. Προχωρούμε σε partnerships με περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς φορείς, αλλά και με όλους τους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όπως την Interpol, την Πικαίο. Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι επίσης το WACI, η African West Coast Initiative, δηλαδή που ε, και εκεί οι εταίροι της συμμετέχουν. Και επίσης το Airport Communication Project που ε, είναι μια συνεταιριστική ας πούμε πάλι προσπάθεια και εμείς νομίζουμε ότι πραγματικά αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα επιτρέψει ε, ακόμα στενότερη συνεργασία και βέβαια και συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη που είναι πάρα πολύ σημαντικά και που ακούστηκαν και προηγουμένως, η ενεργός δηλαδή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, καθώς και πολλών χωρών μελών της. Βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή με εκπροσώπους επιτόπου στην περιοχή. Βέβαια, καλωσορίζουμε τις εξελίξεις αυτές και θέλουμε πολύ να προωθηθούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας απευθύνω αυτά τα λόγια στο σημαντικό φόρουμ που είναι η Επιτροπή σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε έτσι στενότερον στην περιοχή του Σαχέλ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους τρεις σας ε, για αυτές τις εισηγήσεις ε, πληρέστατες ε, παρόλο που είναι ιδιαίτερα ευρύ το θέμα. Διάφορα σχόλια τώρα, ερωτήσεις. Ότι ο Κερκόφε, δεν είναι ότι υποστηρίζει κανείς τον ένα ή τον άλλο εξετάζοντας αυτό το θέμα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς ε, και τους κύριους στόχους καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά συνδυάζονται στενά με την πολιτική ανάπτυξη ε, που έχει για μας την προτεραιότητα. Γι' αυτό, για να μην ξεκινήσει γι' αυτό ένα θέμα, εδώ για την ασφάλεια ασχολούμε, θα είναι ο λόγος υπαρξή μας, αλλά να μην ξεχνάμε την ανάπτυξη. Και ακριβώς ε, η παρουσίασή σας έδειξε τη στενή σχέση αυτών. Ένα ακόμα σημείο τώρα. Ο σφαιρικός χαρακτήρας αυτών των προκλήσεων δύσκολο είναι κανείς να πει ακριβώς από πού ξεκινάνε και πού τελειώνουν οι απειλές. Είπατε για την ε, πυρηνικό τρόμο και προς το παρόν δεν είναι το πραγματικό, αλλά οι χώρες που παράγουν ουράνιο η διάσταση αυτή ίσως ε, υπάρξει και καταλαβαίνετε την ε, ε, το ευρύ φάσμα απειλών που θα μπορούν να προέρχονται από εκεί. Και ακόμα για να απομονώσουμε μόνο το τρομοκρατό εγκληματικό ή το τρομοκρατικό δεν είναι δύσκολο να το ξεχωρίσουμε από τα 10 προβλήματα κάθε κράτους και από το ε, χειροχικό χαρακτήρα που έχει το κάθε κράτος. Ο κ. Μπλάνκο μας είπε για τις πολιτιστικές διαφορές, ας πούμε, στη σύνθεση της Μαυριτανίας ή του Άρεγκα στον Ήγηρα και στο Μαλί. Υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Πολύ δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους για να ασχοληθεί ξεχωριστά και ανάλογα με το κάθε φαινόμενο. Επίσης τη δυσκολία περί περιφερειακής συνεργασίας. Αν δούμε τις τρεις χώρες της Σαχέλ, Μαυριτανία, Μαλή και Νίγερα, στο δεν μπορούμε να δώσουμε εύκολα απαντήσεις χωρίς να λάβουμε υπόψη μας και το ρόλο της Αλγερίας και της Λιβύης και κάτι παραδίπλα. Ε, ξέρετε, με, ακούσαμε για αυτές τις δύο περιοχές κρίσης με διάφορες απειλές που φτάνουν μέχρι και τον κόλπο της Γουινέας. Αναφέραμε και τις πειρατές και την ε, λαθρεμπόριο ε, ναρκωτικών σε συνδυασμό με τον νοτιμαρικανικό λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αυτά λοιπόν και γεωγραφικά έτσι θα πρέπει να εξεταστούν. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τους υπόλοιπους που συμμετέχουν σε διεθνές επίπεδο στην περιοχή αυτή. Τα Συνωμένε Πολιτείε κυρίως που με την προηγούμενη κυβέρνηση, η Προεδρία είχαν μια εταιρική σχέση πάνω σε αυτά ειδική και βλέπαμε όμως ότι ήταν και ιδεολογική η τοποθέτηση γιατί ήταν για την ανδρομοκρατία συγκεντρωμένη λιγότερο στην ανάπτυξη του κόσμου. Τι γίνεται όμως εκεί, τι ακολουθούν, ποιοι είναι οι προσανατολισμοί του σήμερα εκεί εσείς που ξέρετε την περιοχή και ίσως και περιθωριακά, αλλά μιλάμε για το πώς μπαίνει στην Αφρική η Κίνα οικονομικά απέναντι στις ε, οικονομικές αυτές προκλήσεις στην Αφρική. Η Κίνα μπαίνει και αυτή στη μέση ακριβώς το θέμα της ασφάλειας ε, και το πώς μπορούμε κάτι να κάνουμε για τις πρώτες σύλλες ε, γιατί είπαμε αυτές τις τρεις χώρες που έχουν αυτά τα ευαίσθητα προϊόντα ορυκτά, και ακόμα ένα ερώτημα. Πολύ σωστά είπατε κύριε Λόπες Πάγκο ότι απ' έξω προέρχεται ε, η παρέμβαση στην δρομοκρατία και στο Μάλι τελευταία υπενθυμήθηκε ακριβώς ο ρόλος εκείνων που προωθούν προς αυτό από το Πακιστάν και την τρομοκρατική απειλή. Τι γίνεται ακριβώς, ποια είναι η προέλευση εκείνων που συμμετέχουν τώρα ε, στο Μαντράς, Πακιστάν και λοιπά και άλλοι για να ξέρουμε καλύτερα και να δούμε καλύτερα ποια μπορεί να είναι αυτά τα δίκτυα. Αυτά είναι τα δικά μου ερωτήματα, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Νικολάη, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ για τόσα μας είπατε. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν συζητιέται πολύ στην κοινή γνώμη, ούτε καν είναι στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όταν πρόκειται για θέματα διμερεί, όπως είναι οι απαγωγές, οι χώρες αντιδρούν μεμονωμένα, χωρίς να βλέπω να υπάρχει κάποια συνεκτική στρατηγική όσον αφορά την περιοχή του Σαχέλ. Έχω μια ερώτηση που έχει να κάνει με την κατάσταση όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Δεν έχουμε πραγματικά τρομοκρατικά δίκτυα όπως είναι η Ελκαΐδα πρόκειται για εξαγωγή τρομοκρατίας, ναι, αλλά την άλλη μεριά υπάρχουν στην περιοχή οργανώσεις που να είναι τρομοκρατικές ντόπιε ή πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα απ' έξω. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε για την αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει τέτοιες οργανώσεις, είτε το δικαστικό σύστημα, η διακυβέρνηση. Είσαστε αρμόδιος για το θέμα αυτό, συντονιστής μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, για την ανάπτυξη, γιατί για μένα το θέμα της ασφάλειας είναι αυτό που μας καίει σήμερα, αλλά η ανάπτυξη είναι αναγκαία. το μέλλον πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ανάπτυξη όταν ετοιμάζουμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, να γνωρίζουμε όμως προηγουμένως καλά τι συμβαίνει στην περιοχή και έτσι να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μέτρα ανάπτυξης για την περιοχή. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ για όσα είπατε. κατανοητά ιδιαίτερα ήταν και περίχαν πολλά. Και επίσης για το ρόλο της Κίνας και των ΗΠΑ. Θα ήθελα ορισμένα πράγματα να ρωτήσω, γιατί ότι δεν ε, υπάρχει στρατηγική, είτε η Ευρώπη καημένη δεν είναι και τόσο καλά οργανωμένη για να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή στην περιοχή Σαχέλ. Τι γίνεται, τι γίνεται με τα λίτρα. Ορισμένες χώρες δεν πληρώνουν λίτρα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν λίτρα. Τι γίνεται όμως έτσι χρηματοδοτείται η τρομοκρατία. Ταυτόχρονα όμως ε, δείχνει και στοιχεία από προσανατολισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πέστε μας, ε, τι συστήνετε εσείς τα κράτη-μέλη μας ε, για το θέμα αυτό, τι γίνεται με τη χρηματοδότηση με αυτόν τον τρόπο των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Κύριε Ντεκερκόφ, στην αρχή είπατε κάτι ότι και άλλες σειράξεις έχουν ε, σημασία, είναι σπουδές για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αυτές τις απειλές από αυτή την περιοχή και μυρίσατε για τη Δυτική Σαχάρα. Πρόκειται για σύραξη και αντιπαράθεση γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς θα διαλέξαμε να παραστήσουμε το στροθοκαμήλους ε, Η κυρία Φερέρ μου λέει ότι είμαστε διηρημένοι για το θέμα αυτό. Ο κύριο Σολάνα, εντάξει, είπε τι να πω, είναι θέμα των Ηνωμένων Ο καθένα παραπέμπει σε άλλον. Άρα λοιπόν, στρωθοκάμιλοι. Η Αλγερία και το Μαρόκο με κράτη με ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την περιοχή αν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν και με την προέλευση όλου αυτού του προβλήματος ε, και σε αυτά τα θέματα, τότε περισσότερο αποτελεσματικοί θα μπορούσαμε να είμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει για τη βοηθήσει το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας, που από μόνο του προκαλεί αναζωπήρωση του, της τρομοκρατίας. Και παλιότερα εγώ ήμουν μάρτυρας αυτών των γεγονότων παλιά η Λιβύη έχει κάποιο ρόλο, αλλά το Μαρόκο και η Αλγερία αν θα μπορούσαν να συνεργαστούν, τα πράγματα θα άλλαζαν στην περιοχή αυτή ίσως. Και με χώρες που ξέρουμε, όπως το Μαρόκο, που παίρνει βοήθεια για την ανάπτυξη πολλά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ούτε και εξηγεί τι κάνει, πώς περνάνε αυτά τα χρήματα και στον κόσμο της Δυτικής Σαχάρας που είναι στις περιοχές όπου έχει σημειωθεί αυτή, αυτή με τον τρόπο η απεικιοποίηση στον κατάλογο των εθνών. Τι γίνεται και οι Ισλαμιστές και οι Μουσουλμάνοι Στην περιοχή αυτή όμως βλέπουμε ότι κυκλοφορούν ναρκωτικά, λαφρεμπόρο ναρκωτικών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια παρόμοια αποστολή USDP. Όχι όμως σύμφωνα με τις ανάγκες και είναι και θέμα διαχείρισης, διακυβόρυνσης, ε, αναθεώρησης των ρυθμίσεων, να μην αφήσουμε τους ε, πρώην να ασχολούνται με ε, παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες, που το ναρκωτικών, εντρομοκρατία και από ό,τι κατάλαβα την ε, αποστολή SDP την κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι χαζό, δεν, στέκει. Είναι αντίθετο με την κατάλληλη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθεί για να λυθεί το πρόβλημα. Όπω ο κ. Ρούστρομ το είπε και εκεί σημειώνεται αυτή η απειλή μέσω της τρομοκρατίας, μέσω της πειρατείας, όλο και περισσότερο εμφανίζεται αυτό και μήπως θα μπορούσα να μας πει τι γίνεται με την πυρηνική απειλή στην περιοχή αυτή και ο που παράγει ουράνιο, αλλά κάτι το πιο συγκεκριμένο για να δούμε τι γίνεται. Γιατί τώρα και στην Επιτροπή μας θα πρέπει να αποφασίσουμε για το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μάχη κατά της ε, διασποράς των πυρηνικών όπλων, βιολογικών όπλων κλπ. Η κυρία Λεβά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις τόσο πλήρεις παρουσιάσεις σας. Όντως, πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα με πολλές επιπτώσεις. Θέλω να επανέλθω λίγο στο εξής. Η διάσταση της τρομοκρατίας με ποιο τρόπο βρίσκεται παρούσα. Πρόκειται για εγκληματικότητα, σε τι βαθμό και ποια είναι η σχέση των δύο μεταξύ τους. Γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είδαμε στο Αφγανιστάν και αλλού τι γίνεται όταν έχουμε τρομοκρατία καταλήγουμε σε πράγματα και σε δράσεις οι οποίες τελικά δεν ξεριζώνουν την αιτία. Γίνονται διαφορετικές αξιολογήσεις, πολύ μάλιστα διαφορετικές μεταξύ τους κάθε φορά που μιλάμε για την πυρηνική τρομοκρατία, για παράδειγμα, έτσι κι νομίζω ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα προς το παρόν. Έπειτα για τις συγκρούσεις με το Μαλί και στο Μαλί και αυτά είναι πράγματα πολύ παλιά. Δεν μπορεί να υπάρχει στρατιωτική λύση. Μιλήσαμε για στρατιωτικές βάσεις στο Βόρειο Μαλί. Βάσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες στον κόσμο. Για μένα οι βάσεις αυτές θεωρούνται από τον κόσμο σαν κατοχικές δυνάμεις και κάνουν τελικά το πρόβλημα οξύτερο. Υπάρχει και το πρόβλημα της ε, συμμετοχής των Αμερικανών, των Ηνωμένων Πολιτειών. 100.000 δολάρια θα δίνονται μάλλον κάθε χρόνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο Μαλί. Και ορισμένοι λένε ότι ακόμα και τα χρήματα αυτά τελικά έχουν σαν αποτέλεσμα η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα για να καταπολεμήσει το έγκλημα. Γιατί μόνο όσο υπάρχει εγκληματικότητα θα συνεχίζουν να φτάνουν τα χρήματα αυτά στην κυβέρνηση του Μαλή, η οποία τα χρησιμοποιεί και για άλλους λόγους που δεν έχουν ε, πάντα άμεση σχέση με τον αρχικό λόγο και αιτία για την οποία στέλνονται τα χρήματα αυτά στο Μαλή. Είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Εσείς αναφερθήκατε στην κατάρτιση και πόσο σημαντική είναι στα πλαίσια της τρομοκρατίας. Υπάρχει αναλφαβητισμός τεράστιος στις χώρες αυτές. Δεν φταίει η τρομοκρατία. Το ποσοστό των αναλφάβητων υπάρχει και δεν φταίει η τρομοκρατία γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω και επιμένω ότι πρέπει να γίνονται επενδύσεις στην εκπαίδευση Μάλιστα το Μαλί είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Και ούτε και σε αυτό φταίει η τρομοκρατία. Αλλά φταίνε ένα σωρό άλλοι παράγοντες οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ το πλαίσιο της σημερινής μας συζήτησης. Πρόκειται για αιτίες που έτσι καλώ δεν θα λυθούν σήμερα. Έχω όμως μια ερώτηση για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Εσείς αναφέρατε προγράμματα στήριξης σε διάφορες χώρες. Προσπάθησα εγώ να μάθω και τελικά δεν ξέρω ποιο είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών στην περιοχή του Σαχέλ. Μας μιλήσατε για ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πρόγραμμα. Και έπειτα αναφερθήκατε σε αύξηση των πιστώσεων. Θέλω να ξέρω πώς βλέπετε εσείς ακριβώς τα πράγματα. Και έπειτα η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε στην πληρωμή ή μη πληρωμή λίτρων. Κύριε Κερκόβ, είπατε ότι αιτιολογείται το να πληρώνει κανείς λίτρα. Τουλάχιστον στις 10 Σεπτεμβρίου, αυτό είπατε, ε, σε κάποιο site το διάβασα. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε ότι όντως έτσι είναι. Στο μέλλον θα κληθούμε να ελευθερώσουμε ο Μύρους ξανά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ασχοληθεί. Και εφόσον ναι, πώς είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας και μετά θα ακούσουμε άλλες παρεμβάσεις από τους ευρωβουλευτές. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Και οι συνάδελφοι θα συμπληρώσουν για την Αμερικανική πρωτοβουλία τώρα. Έχουμε μια εξέλιξη εκεί. Με, από τον πρόεδρο Μπούς ε, προσπάθεια ήταν κυρίως αποκλειστικά σχεδόν στρατιωτική και για την στρατιωτική εκπαίδευση και με την πρωτοβουλία της Γαλλίας είχαμε ένα συντονισμό όμως τώρα με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση παντού όλοι και όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη και η προσέγγιση να είναι κυρίως του τύπου του ευρωπαϊκού. Να λοιπόν που αλλάζουν τα πράγματα και αντιλαμβανόμαστε από κοινού την ε, απειλή και θέλουμε όλοι μια κοινή πολιτική ολοκληρωμένη, σφαιρική. Και εντάξει, δεν θέλουμε τώρα να στραβωθούν τα πράγματα, αλλά υπάρχει περισσότερες αποχρώσεις στην αντιμετώπιση των Αμερικανών ε, και για την Κίνα, τι να σας πω τώρα δεν είδα κινέζικη παρουσία τόσο δραστήρια, τουλάχιστον όπως στο Κονγκό ή στην Κεντρική Αφρική, που εκεί υπάρχει παρουσία κινέζικη, αλλά για ιστορικούς λόγους, για σιδερούχες ενώσεις για τη Μαυριτανία και ουράνιο για τον Ήγερα. Προς το παρόν όμως οι υπόλοιποι είναι στραμμένοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, προς ορισμένα κρατημέλη. Και ακόμα κάτι. Ορισμένοι που παροτρύνουν προς μια κατεύθυνση αρνητική ε, είναι Πακιστανοί και η Σαουδική Αραβία στη Μαυριτανία όμως. Ε, και δεν είναι ένδειξη, εντάξει, μη μου ε, με ερμηνεύσετε λανθασμένα. πάρα πολλά κρέα τζαμιά τα τελευταία, τελευταία δέκα χρόνια και επίσης ε, στη Μαυριτανία για την κατάρτιση ε, δικαστών βάσει της Σαρία ε, του Ισλαμικού νόμου και αντί για κλασική προσέγγιση ποινική σημαντικά πρότυπα και η κατάσταση κυρίω στη Μαυριτανία αυτό μα είχε και όπω είπε Μανουέλ στο νότο του Νίγηρα και με την επιρροή της Νιγηρίας στα βόρεια αλλά σίγουρα υπάρχει αυτό ο προσελκυσμό και θα πρέπει να τον προσέξουμε. Η κυρία Νικολάη αυτό που ρώτησε. Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε μια στρατηγική όπως ε, είπαμε να λάβει υπόψη της αυτοδεγική όλες τις πτυχές του οργανωμένου εγκλήματος. Τι γίνεται τώρα με τα λίτρα που είπαν η κυρία Γκόμενς και Λέζιν ότι δεν υπάρχει μια σαφή συγκεκριμένη και οργανωμένη εικόνα πάνω σε αυτό. Όχι, ναι. Και να σου το πω καθαρά. Δεν νομίζω να πω ότι είμαι υπέρ της πληρωμής λίτρων, το αντίθετο είχα πει και σίγουρα η πληρωμή δεν είναι κάτι το θετικό. Η Αλγερία έθιξε ιδιαίτερα το θέμα αυτό πέρυσι και φέτος. Ήμουν στην Γενική Συνέλευση των Εθνών τη βδομάδα που μας πέρασε και το προβάλλει αυτό το θέμα η Αλγερία από τη Συμβοσφαλίας και από τη Γενική Συνέλευση θέλει να υιοθετηθεί ένα ψήφισμα για το 1904 ψήφισμα με μια τη σκέψη ότι ναι, είναι έτσι περνάνε τα χρήματα στην δημοκρατία και να συμπληρωθούν αυτά οι ρυθμίσεις των ΕΕ για την δημοκρατία και με μια συγκεκριμένη αναφορά για το θέμα αυτό. Τώρα παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα επηρεάζει την κατάσταση στην περιοχή και επαναλαμβάνω δεν είναι θετικό να πληρώνονται λίτρα και στην παρέμβασή του στους πρέσβεις 26 Αυγούστου μας πέρασε ο πρόεδρος Σαρκοζή είπε ότι δεν θα πρέπει απλά και μόνο να πληρώνουμε λίτρα αυτή να είναι η στρατηγική μας αυτήν υιοθετούμε και έτσι να ελεύθερονται όμοιροι και βοήθησε φεβελία και στην απελευθέρωση στο Μαλί ομήρων και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα πάνω σε αυτά. Για τη Δυτική Σαχάρα τώρα, εντάξει, εμείς απαντά τα ίδια πράγματα όπως και η Επίτροπος Φερέρο και ο Σολάνα. Μη σε παραλαμβάνω τα ίδια, αλλά το είπαμε, εντάξει, δεν είμαι ειδικό πάνω σε αυτό, γι' αυτό θα προσέξω να μην κάνω σχόλια σε τόσο περίπλοκα θέματα, αλλά μας απογοητεύει όλα αυτά, γιατί το Μαρόκο δεν μπορεί να βοηθήσει, γιατί δεν μιλούνται οι δύο χώρες, είναι κλειστά τα σύνορά τους και χρειαζόμαστε και την Αλγερία και το Μαρόκο ε, δεν θα τεθεί μια λύση εκεί χωρίς να συμμετάσχει ιδιαίτερα η Αλγερία που είναι σημαντικός παράγων εκεί και το Μαρόκο όπως και η Μαυριτανία και καταλαβαίνετε ότι είναι και μεγάλη δυσκολία του θέματος ε, και στο average για το Μαρόκο Ναι, δίνουμε 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο όπως στο Μαλί και υπάρχει μια ενισχυμένη εταιρική σχέση με το Μαρόκο έτσι γιατί η Γουινέα Μπισάου θα αφήσω τη συναδέλφου συναδέλφους που γνωρίζουν καλύτερα το θέμα από μένα αλλά κρίμα που αποσυρθήκαμε από εκεί και για τους λόγους ε, που αποσυρθήκαμε για το Αφγανιστάν μέχρι την Γουινέα Μπισάου, αν δούμε αυτές οι αποστολές ε, πέρα από αυτό είναι προς, την, ε, προς το κέρας Αφρικής οι αποστολές μας και προς τα δυτικά δεν έχουμε, δεν υπάρχουν αποστολές δικές μας. Θα πρέπει να το αναρωτηθούμε αυτό, τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων Άστον, ασχολείται με αυτό. Μερικές φορές ξεκινώντας μια αποστολή δεν αναρωτιέται και το τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα περατώσει την αποστολή της. Θα πρέπει να έχουμε εργαλεία μέσα λεπτότερα και όχι μόνο εντάξει τρεις τεχνικοί σύμβουλοι... να πάνε εκεί στην αντιπροσωπεία στον Παμακό. Τι γίνεται, τι σημασία έχει, ή να βάλουμε 50 στρατιωτικούς εκεί. Θα πρέπει να δούμε πιο λεπτά μέσα και στην άλλη βασικότητα με αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε 20 άτομα. Ε, μια αποστολή περιλαμβάνει πολλά μέλη, κοστίζει κλπ. Μήπως θα μπορούμε να έχουμε μέσα πιο ευέλικτα, αλλά για το ΣΕΧΕΛ εκεί θα πρέπει να το εξετάσουμε, να το συζητήσουμε το θέμα. Και ήταν και από τα τελικά που ερώτησα για το Μαλί γιατί στο Βόρειο Μαλί για να έχουμε και πάλι την παρουσία του κράτους, να έχουμε στην δικαιοσύνη, στην ασφάλεια, στην διοίκηση, τι γίνεται ε, από τον Παμακό. Μπορεί να γίνει, ίσως χρειάζονται 150 άτομα, να δούμε ένα ελαφρότερο, πιο ευελικτό μέσο. Κύριε Λεζένιο τρομοκρατία ή οργανωμένο έγκλημα. Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι τρομοκρατία. Το ζήσπεση το... της Αλγερίας είναι η ακμή. που στην Αλγερία είχε κάπως καταπιεστεί και αναζωπηρώθηκε και με την Αλκάιδα δεν νομίζω να υπάρχει άμεση κοινό έλεγχο και χρηματοδότηση αλλά ο, τα λόγια που χρησιμοποιούν και τις ε, απόπειρε απόπειρες καμικάζι και στον ΟΗΕ και σε επίσημα κτίρια κλπ. Έτσι το GSPC και πάλι πήρε ένα καινούριο ρόλο και προσέλαβε και καινούρια μέλη ίσως μπαίνει στη μέση και η, μαφία, καταλήγει σε μαφιόζικες ενέργειες. Οι ΦΑΡΚ στην Κολομβία καταλήξαν ε, μαφιόζοι, παράγουν και πουλούν ναρκωτικά. Και σε άλλες περιοχές του κόσμου δυστυχώς έτσι γίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα η ακμή πόσο συμμετέχει στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και στα διάφορα λαθρεμπόρια. Από σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το διαφορετικό, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Υπάρχει και η διάσταση ιδεολογική, έτσι, να μην περασυρώμαστε. Δεν μιλάμε για αερασβαστικό νέο χαρακτήρα στο Ιγέρα. Δεν είναι μόνο ότι ψάχνουν για κέρδος χρήματα. Αυτό λοιπόν ιδιαίτερα θα πρέπει να μας ανησυχεί. Ότι δίνουν 100 ε, εκατομμύρια ευρώ Αμερικάνοι. Ε, όχι, όχι, δεν με ανησυχεί αυτό. Νομίζω ότι είναι παίζει παθητικό ρόλο το Μαλί επειδή παίρνει χρήματα. Αντίθετα, πείθεται ότι θα πρέπει να δει κανεί καθαρά ποιε είναι οι απειλέ και το είπε και συναδελφοί. Με τον πρόεδρο του Μαλί συναντήκα δύο φορέ και περισσότερο μου μίλησε για το Στουαρέγ παρά την ΑΚΜΗ την πρώτη φορά ο πρόεδρο του Μαλί. Τη δεύτερη φορά τον Ιούλιο στη συνάντηση δεν ήμουν παρόν, αλλά νομίζω ότι ακούστηκε εκεί, το άκουσαν και άλλοι και έκανε μια παρουσίαση πραγματικής στρατηγικής ε, του Μαλή. Θα πρέπει να του συμπαρασταθούμε και πρότεινα την αντιπροσωπεία των Μπαμακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να χαράξουν ένα οδικό χάρτη και να βλέπουμε τις διάφορες φάσεις ε, του σχεδίου Πυρήν και με τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Μαλή. Γιατί θα φτιάξουμε τώρα, κατασκευάσουμε δρόμους, θα προσφέρουμε χρήματα, αν δεν υπάρχει διάθεση μόνιμη από τις αρχές του Μαλή να επενδύσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα ο πρόεδρος και η κυβέρνηση του Μαλή κατάλαβαν ποιο είναι το πρόβλημα και θα πρέπει και εμείς τώρα να το συμπρασταθούμε. Και η κατάρτιση θα πρέπει να προσπαθήσουμε, δεν τα ξεκαθάρισα κιόλα, ότι χρειάζεται ε, όχι μια μόνο προσέγγιση για την ασφάλεια που τα απετύχανε. Τώρα εντάξει να πάμε στρατιωτικού εκεί χωροφύλακε, τώρα το άλλο αν δεν ασχοληθούμε με την Κίνταλγκάο και άλλε περιοχέ ε, στο βόρειο του Μαλί και στο ε, ρισπαστικό χαρακτήρα περί το Μαλί και όλα αυτά τα πράγματα να ασχοληθούμε με αυτά και όλα τα προβλήματα αλλά να είναι ειδικοί πάνω σε αυτά τα θέματα για τις ε, νομαδικές φυλές όλα αυτά είναι πράγματα που θα μπορούσαν να επανεξεταστούν ε, σε αυτό το μέρος του Σαχέλ. Είμαι πεπισμένο και εγώ όπως και εσείς ότι η εκπαίδευση είναι πολύ βασικό στοιχείο. Δεν είναι επειδή είμαστε αναλφάβητοι που γινόμαστε τρομοκράτες, αλλά σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό, σε αυτό που ονομάζουν ε, στον ΟΗΕ την αιτία που βοηθάει στο να αυξάνεται η δρομοκρατία. Φυσικά δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε αμόρφωτοι γινόμαστε δρομοκράτες, όχι. Αν όμως είμαστε μορφωμένοι, ε, μειώνονται οι πιθανότητες να οδηγηθούμε στην τρομοκρατία. Δεν βλέπετε καθαρά το τι έχει αποφασιστεί επειδή είμαστε στο στάδιο των επιλογών. Ε, βραχυπρόθεσμα πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις, αλλά μακροπρόθεσμα είμαστε σε μια βούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προχωρήσουμε. Ευχαρίστως πάντως να σας στείλουμε ό,τι στοιχεία έχουμε για τόσα έχουν ήδη αποφασιστεί και αυτά τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της απόφασης, χωρίς να έχουμε καταλήξει ακόμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ από την πλευρά μου θα επικεντρωθώ στο θέμα της συνεκτικής στρατηγικής, γιατί είναι κάτι που επανέρχεται κάθε τόσο. Αυτό ακριβώ προσπαθούμε να πετύχουμε, να δώσουμε συνοχή σε μια στρατηγική που φτιάχνουμε. Γιατί είναι αλήθεια ότι αρχικά δεν υπήρχε. Αν υπήρχε αυτή η συνοχή, δεν θα χρειαζόταν να την ψάξουμε. Αναγνωρίζουμε συνεπώς, αυτή είναι η απόψή μου τουλάχιστον, ότι δεν έχουμε ακόμα μια συνεκτική στρατηγική για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αν την είχαμε, θα είχαμε προχωρήσει πολύ. Όμως κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για να υπάρξει μια τέτοια στρατηγική στο τραπέζι του Συμβουλίου. Με δράσεις, ορισμένες από τις οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν προγράμματα που έχουν ξεκινήσει. Στην ερώτηση της κυρίας Νικολάη, που επίσης έρχεται και ξανάρχεται, τα μέτρα ανάπτυξης. Τι μέτρα ανάπτυξης έχουμε. Και η κυρία όχι στρατιωτικές λύσεις είπατε. Και ότι οι βάσεις είναι σαν δυνάμεις κατοχής στο Βόρειο Μαλί, ότι έτσι τις νιώθει ο κόσμος. Μα ακριβώς έτσι φτάνουμε και στην καρδιά του προβλήματος. Δηλαδή πώς να βοηθήσουμε με εκπαίδευση σε έναν χώρο όπου οι δάσκαλοι, οι καθηγητές είναι θύματα επιθέσεων. Χωρίς ασφάλεια δεν μπορούμε να έχουμε εκπαίδευση. Χωρίς ασφάλεια δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ανάπτυξη, ούτε εκπαίδευση. Είναι ο φαύλος κύκλος που έλεγα και πριν. Πώς αυτός ο φαύλος κύκλος θα γίνει ένας καλός κύκλος, ένας θετικός, έτσι ώστε να τροφοδοτούμε το καλό αντί για το κακό. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ορθή στρατηγική από την κυβέρνηση του Μαλή για να ξαναπάρει τον ε, Βορρά. Να τον πάρει, ναι, αλλά από ποιον. Το θέμα είναι να μην δημιουργηθεί νέα αιστεία σύγκρουσης. Σίγουρα όμως πρέπει το κράτο να ξαναβρεθεί στο Βορρά. Γιατί τελείω ποιο θα φροντίσει για την εκπαίδευση εκεί, ποιο θα φροντίσει να υπάρχουν ε, κοινωνικέ ε, παροχέ και υπηρεσίε, ποιο θα δημιουργήσει απασχόληση. Μόνο το κράτο μπορεί να το κάνει αυτό. Αν το κράτο είναι απόν από το Βορρά, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που θα το κάνουν γιατί δεν είναι παρούσε εκεί, γιατί φοβούνται, μην απαχθούν, υπάρχει κενό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πώς θα συνοδεύσουμε την παρουσία του κράτους έτσι ώστε να νιώσει ασφάλεια και να έχουμε στη συνέχεια μία δράση υπέρ της εκπαίδευσης, υπέρ της συμφιλίωσης. Να νιώσουν τα θετικά από την ειρήνη οι άνθρωποι στην περιοχή. Ένα από τα πρώτα προβλήματα λοιπόν που μας υπογράμμισαν οι του ΑΡΕΚ είναι η απομόνωση. Ότι δεν υπάρχουν ε, δρόμοι, δεν υπάρχει τρόπος. Στο Κιντάλ οι αγορές έχουν τις προμήθειές τους από την Αλγερία και όχι από την υπόλοιπη χώρα. Τα εμπορεύματα έρχονται από την Αλγερία ή από τη Λιβύη στο Κιντάλ και όχι από τον Παμάκο. Άρα η περιοχή αυτή της χώρας οικονομικά είναι περισσότερο συνδεδεμένη με τις βόρειες χώρες παρά με την ίδια χώρα. Υπάρχει η προσπάθεια λοιπόν σύνδεσης μέχρι το Κιντάλ. Το δρόμο αυτό που να συνδέει την πρωτεύουσα με το Κιντάλ είναι κάτι που όλοι το ζητάνε, γιατί προσφέρει και ευκαιρίες για απασχόληση. Τώρα, ποιες είναι οι στρατηγικές ανάπτυξης. Πρώτον, ενίσχυση της χώρας, ε, του κράτους μάλλον πιο συγκεκριμένα, του κράτου, ώστε το κράτος να μπορεί να προσφέρει την ασφάλεια και όπως είπε και ο συνάδελφο, με τρόπο που ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι η δικαιοσύνη, ο νόμος, η αστυνομία, όλα αυτά να εντάσσονται μέσα στην στρατηγική μας που να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, να τα βλέπει θετικά. Συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΑ πολύ. Και ποιος είναι και ο ρόλος του στρατού, γιατί και ο στρατός εννοείται ότι έχει γνώση για αυτά τα ζητήματα και μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Για την Γουινέ Μπισάου τώρα που με ρωτήσατε, που υπάρχει το πρόβλημα της αποστολής ΣΔΠ. Ολοκληρώθηκε η αποστολή. Η αποστολή ήταν το νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση του κράτους και πώς το νομοθετικό πακέτο θα γίνει επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το Κοινοβούλιο το ψήφισε το πακέτο, αλλά η Προεδρία δεν το πρόθεσε ακόμα. Τα επόμενα στάδια είναι πολιτικής φύσεως. Θα μπορούσε η αποστολή να έχει συνεχιστεί για λίγο, για να βοηθήσει στην εφαρμογή. Αλλά πολιτικά υπάρχει μπλοκάρισμα υπάρχει κάτι σαν πραξικόπημα που δεν λέγεται έτσι μεν, αλλά λίγο πολύ είναι κάτι τέτοιο, ότι οι στρατιωτικοί παίρνουν την εξουσία. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση όπου πιέζουμε πολιτικά, ώστε η πολιτική, πολιτικο-στρατιωτική τάξη στη Γουινέα Μπισά, διακόπτει η κυρία Γκόμες εκτός μικροφώνου, απαντάει ο κύριος Μπλάνκο, πάντως οι υπηρεσίες του Συμβουλίου αυτή την εποχή προσπαθούν να δούνε πώς μπορούν να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με τη Γουινέα Μπισάου. Αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Είναι μια δυνατότητα. Μια που υπάρχει μια πολιτική μετάβαση που οδηγεί σε οπισθοχώρηση. Δηλαδή χάνεται το κεκτημένο σε ένα μεγάλο βαθμό και είναι κρίμα. Για το ποσοστό αναλφαβητισμού, ναι, πρέπει να βοηθήσουμε την ανάπτυξη, τη μόρφωση και να μην θυσιάσουμε τίποτα. Αλλά μια χώρα η οποία είναι τόσο εύθραυστη, τόσο ευάλωτη εξαιτία τη διαφθορά, εξαιτία τη ακμή, εξαιτία του λαθρεμπορίου, καταλαβαίνετε ότι το κράτο δεν έχει πολλές δυνατότητες να προσφέρει κοινωνικά μειώνονται οι δυνατότητες του. Γι' αυτό και χρειάζεται μια στρατηγική που να καλύπτει και την ανάπτυξη και την ασφάλεια. Αυτά τα δύο πάνε μαζί στην περίπτωση τέτοιων εύθραυστων χωρών. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, let me... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρθω πρώτα στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και στο τι απαιτείται κατά την άποψη των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκα ήδη στην συνολική στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών κατά της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε το 2006 και που στον πρώτο της πυλώνα ασχολείται με τις συνθήκες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη τρομοκρατίας καθώς επίσης με θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Κράτος δικαίου εντάσσεται μέσα σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής η οποία να μπορεί πράγματι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των χωρών. Στα πλαίσια αυτά η εκπαίδευση βέβαια είναι ένα σημαντικό θέμα. Η UNESCO είναι ένας από τους 30 φορείς των Ηνωμένων Εθνών που είναι, συμμετέχουν σε αυτή την ε, ε, task force και μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών βέβαια, η περιοχή του Σαχέλ είναι μια περιοχή η οποία θεωρήθηκε εξ αρχής ότι θα πρέπει να επωφεληθεί από τη συλλογική δράση CTRF που έχει ήδη αποφασιστεί να, να ε, μπει σε ενέργεια για την καταπολέμηση γενικά του αλφάβητισμού, για παράδειγμα. Πιστεύουμε πάντως ότι χρειάζεται ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης βασισμένο σε κράτος, σε δικαίου και με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως μόνη πραγματικά αποτελεσματική δράση κατά της τρομοκρατίας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό στις χώρες αυτές να εξασφαλίσουμε ώστε όσοι ασκούν την ποινική δικαιοσύνη να χαίρουν της απαραίτητης εκπαίδευσης. Τέθηκε το ερώτημα, για παράδειγμα, τι, πώς ορίζεται η κλιματικότητα και πώς ορίζεται η τρομοκρατία. Μπορούν να είναι ταυτόχρονα ε, ενέργειες εγκληματικές και ενέργειες τρομοκρατικές. Αλλά το γεγονός ότι μόνο μία χώρα στην περιοχή έχει καταφέρει να ολοκληρώσει μία ποινική υπόθεση τρομοκρατικού χαρακτήρα ενώπιον της ποινική δικαιοσύνης δείχνει ότι το ποινικό σύστημα είναι ακόμα ε, εξαιρετικά ασθενές. Δεν ανταποκρίνεται δηλαδή στις ανάγκες που σημειώνονται στον τομέα της ποινική δικαιοσύνης. Όταν τίθεται θέμα ποιες ε, δράσεις είναι τρομοκρατικές και ποιες όχι, οι μόνες ε, τρομοκρατικές ομάδες που θεωρεί ομάδες ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι αυτές του καθεστώτος 627. Και εμείς μιλούμε τώρα για τρομοκρατικές δράσεις οι οποίες δηλαδή πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια των ε, διεθνών εγγράφων, των διεθνών δηλαδή συμφωνιών και ούτω καθεξής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταστήσουμε, να φέρουμε σε θέση δηλαδή όλους όσοι δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της άσκησης της ποινική δικαιοσύνης να ασκούν την ποινική δικαιοσύνη βασισμένη στα ε, έγγραφα αυτά, στα κείμενα αυτά ο ίδιος ο Οργανισμός Εθνών δεν προβαίνει σε ανάλυση των απειλών. Εμείς έχουμε ε, την εντολή να το κάνουμε αυτό για το οργανωμένο έγκλημα. Και από τη σκοπιά αυτή έχει ρηχθεί ιδιαίτερη προσπάθεια στην συλλογή δεδομένων για ε, διάφορες εγκληματικές ενέργειες καθώς και παράνομα εμπόρια στην περιοχή της ΑΧΕΛ. Η έρευνα γίνεται από τη σκοπιά του οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή της καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών. Υπάρχει όμως μια διασύνδεση, όπως γνωρίζουμε, τακτικού χαρακτήρα μεταξύ της Αλκάιδα στο Μαγκρέμπ και εγκληματικών ομάδων. Για την ώρα όμως δεν υπάρχουν ε, σκληρές ενδείξεις, δηλαδή πολύ ξεκάθαρες ενδείξεις, αδιαμφισβήτητες ενδείξεις για περισσότερα ε, πράγματα σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία. Τώρα για την πυρητική τρομοκρατία δεν ασχολήθηκα πολύ, δεν θα, αν ούτε στις ίδιες τις ε, διότι δεν ε, περιλαμβάνονται στην εντολή μα και διότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι συνεργάζονται με εμά και έχουν το καθήκον αυτό και άλλωστε πολλές εκ των χωρών μελών της ε, Ένωσης έχουν την ικανότητα να αναλύσουν την ε, απειλή αυτή. Για, την, για τον Ήγηρα αναφέρατε βεβαίως η Γκάνα επίσης έχει πυρηνικό υλικό στο εδαφός της. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε την ανάλυση από την σκοπιά του δικαίου. Και από αυτή τη σκοπιά είναι ξεκάθαρο ότι κάθε ε, τρομοκρατική ενέργεια η οποία έχει ε, σχέση με πυροβιταχή είναι περιλαμβάνεται δηλαδή στην σκοπιά αυτή της ανάγκης να αναπτυχθούν δράσεις για να αντιμετωπίζονται τέτοιες ενδεχόμενες εγκληματικές ενέργειες. Σε ό,τι αφορά τα λίτρα, θέλω και εγώ να τονίσω ότι βέβαια από τη σκοπιά των Ενωμένων Εθνών και και το ψήφισμα 904 που ανέφερε ο Ζιλ προηγουμένως, η καταβολή λίτρων σε καταχωρημένες ομάδες, στους ε, καταλόγους δηλαδή των ΗΠΑ, είναι παράνομη. Αυτό είναι μία βάση. Τώρα, πέραν αυτού, στις ε, νομικές συμβάσεις που έχουμε δεν αναφέρεται το θέμα των λίτρων. Και τέλος, ένα σχόλιο σχετικά με την προσέγγιση των ΗΠΑ που είναι βέβαια σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή του Σαχέλ. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι στα πλαίσια μιας νέας και πιο ενεργούς στρατηγικής που διατυπάθηκε από την σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να υπάρχει η θέληση συνεργασίας και με πολυμερείς οργανισμούς όπως τα Ενωμένα Έθνη με συνάντηση η οποία έγινε ήδη τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους με όλους τους εκπροσώπους ε, των οργανισμών των Ενωμένων Εθνών και με αμερικανικούς ε, φορείς σε μια προσπάθεια έντασης, εντατικοποίησης του διαλόγου. Βέβαια, και στο πλαίσιο του G8 οι Ενωμένε Πολιτείε, συμφώνησαν να δώσουν υψηλή προτεραιότητα την καταπολέμηση τρομοκρατίας στην περιοχή Σαχέλ και σε στενή συνεργασία με τους φορείς του συστήματος των Ενωμένων Εθνών. Στα πλαίσια της ε, πρωτοβουλίας αυτής της CITF, ε, των, της αντιμετώπισης δηλαδή των θεμάτων αυτών στην περιοχή. Μπένα Ραμπατού. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Αντιστοιχούν σε μία ε, ανάλυση που συμμερίζομαι για το πρόβλημα του Σαχέλ. Η τρομοκρατία στο Σαχέλ ε, δεν είναι κάτι που παρουσιάζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ε, έχει να κάνει με τη φτώχεια των κατοίκων εκεί. Η ΕΚΜΗ δεν προέρχεται από εκεί, αλλά ανταποκρίνονται εκεί γιατί είναι άνεργος ο κόσμος, είναι φτωχός. Είναι αμόρφωτος ή σχεδόν η Ευρώπη, στην Ευρώπη μιλήσαμε πολύ για την προσέγγιση των ΗΠΑ, συμφωνώ. Αλλά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένας ιδιαίτερος εταίρος. Η Αφρική, το Μαγκρέμπ είναι ορίζοντας ε, της, ε, που θα πρέπει προς τα εκεί να η Ευρώπη. Ένας πόλος ε, εντάξει τώρα πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μεσόγειο, αλλά το σκεφτόμαστε αυτό. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται να χάσουμε αυτό το στόχο για την εταιρική σχέση. Δύο άξονες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όχι πια τόση φτώχεια, γιατί αν δεν έχει οράματα και μέλλον ε, η νεολαία, τότε θα περιμένει χρηματοδότηση από τους τρομοκράτες. Δεύτερο τώρα, και πώς θα βαστεί κανείς τα πολιτιστικά στοιχεία εκεί της περιοχής. Από πολλά, πολύ παλιά οι Τουαρέγ διαθέτουν μια κουλτούρα πολιτιστικά στοιχεία. Δεν μιλήσαμε για τη σημασία που έχουν οι γυναίκες εκεί για την εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο το σχολείο που εκπαιδεύεται κανείς. Οι ίδιες οι γυναίκες εκείνες μεταβιβάζουν τα μηνύματα και θα μπορούσαν να δώσουν νέες ιδέες για το, στον κόσμο αυτό με τα πολιτικά στοιχεία τα ομανιστικά και μέσα σε ένα Ισλάμ ε, προσανατολισμένο προς την θεωρία Σούφη ανοιχτό. Και μιλήσατε για τα διαφορά κράτη, ένα ισχυρό κράτο. Σημαντικό είναι βέβαια για μια προσέγγιση σχετικά με την ασφάλεια, αλλά όχι μόνο με τα πολιτιστικά στοιχεία επίση και με την εκπαίδευση. Δεν μιλήσαμε για τους τοπικούς φορεί. Οι ηγέτε των ΑΡΕΓ στις περιφέρειες εκεί, οι τοπικοί φορεί πέρα από τα κράτη μπορούν να βοηθήσουν, είναι επιτόπου, γνωρίζουν το λαό, μπορούν να παίξουν ένα βασικό ρόλο γιατί οι ενέργεια τους ακριβώς κολλάνε στην αντίληψη του εκεί λαού. Εντάξει, εμείς μπορούμε να πούμε εμείς από την Ευρώπη, εμείς θα φτιάξουμε, θα κάνουμε, θα καταρτήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, καλό είναι το κράτος δικαίου, αλλά θα πρέπει εκεί, επί τόπου να μπορεί κανείς να συντροφεύσει, να συνοδεύσει εκείνους που επιτόπου βρίσκονται, κυρίως τοπικούς φορούς, τους ε, περιφερειάρχες, ε, τους ηγέτες των φυλών, ε, για να ξεριζώσουμε το φαινόμενο αυτό της τρομοκρατίας. Κάτι ακόμα και ολοκληρώνω για την κυκλοφορία των πολιτών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν εκεί. Δεν μπορούμε να πετύχουμε μια ένωση και να έχουμε μια εταιρική σχέση και μετά η πολιτική μας να είναι τέτοια που οι νέοι, πώς να το πω να είναι δέσμοι στις χώρες τους, ε, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν. Έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο, έχουμε το καθήκον αυτό στον κόσμο αυτό να υπάρχει μια ιδιαίτερη ε, δυνατότητα κίνησης ε, και να προσέχουμε την πολιτική του ασύλου και ε, την πολιτική για βίζα. Όλα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν. Α, κάτι, κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο. Για το ρόλο της Αλγερίας. Το κουτί της Πανδώρας είναι για την τρομοκρατία. Εκεί άνοιξε το κουτί αυτό. και η πολιτική που ασκήθηκε εκεί είχε τρομερές επιπτώσεις γιατί δεν κατέληξαν δικαιοσύνη οι ένοχοι, οι υποτιθέμενοι ένοχοι. Τα κατάφεραν, βγήκαν και βγήκαν και βρήκαν και δουλειά και τους βλέπουν οι ε, συγγενείς των θυμάτων να είναι ισχυροί κοινωνικά και καταλαβαίνετε και οι υπόλοιποι λένε ε, σκέφτονται «Α, άρα λοιπόν μπορεί κανείς να είναι και τρομοκράτης και να έχει μια ωραία θέση στην κοινωνία στη συνέχεια». Αυτό λοιπόν την κοινωνία να την αποφύγουμε που είναι τρομοκράτες που δεν ε, καταδικάστηκαν και θύματα ή συγγενείς θυμάτων που δεν βλέπουν να απονέμεται δικαιοσύνη. Και το θέμα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αυτό θα πρέπει να έχει μια τρομερά στερεβάση και θα πρέπει να δούμε στην Ευρώπη εσείς ε, τι κάνετε σχετικά με τις χώρες αυτές για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρία Λούνατσεκ. Ε, Ευχαριστώ. Με ενδιαφέρουν θέματα συντονισμού, χρηματοδότησης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτη ερώτηση ο συντονισμός, η συνεργασία ή ο ρόλος τέλος πάντων της Αφρικανικής Ένωσης. Τι συνεργασία υπάρχει. Επίσης, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει την περιφερική συνεργασία. Γνωρίζουμε ότι χώρες όπως η Μαυριτανία, η Αλγερία ακολουθούν ή θέλουν να ακολουθήσουν περισσότερο μια επιθετική ε, στρατιωτική στρατηγική, ενώ το Μάλι λιγότερο. Πώς μπορούν να συντονιστούν λοιπόν οι στρατηγικές τους και τελικά ποια στρατηγική θα επιλεχθεί εάν δεν επιτευχθεί αυτή η συνένεση. Επίσης, η Κομισιόν χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, και εκπαίδευση αστυνομικών δυνάμεων και δικαιοσύνης. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι πώς εκπαιδεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Πρώτον, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν ταχαίως ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και δεύτερον για να μην προβαίνουν σε τέτοιες παραβιάσεις και οι ίδιοι. Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ για τον μηχανισμό αυτών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των γυναικών, πώς είναι δυνατόν, πώς γίνονται λοιπόν σεβαστά αυτά, ώστε το προσωπικό αυτό το οποίο ε, υφίσταται την εκπαίδευση να μην προβαίνει σε τέτοιες παραβιάσεις ανθρώπινων και άλλων δικαιωμάτων. Κύριε σε αυτό που ρωτήσατε για το ρόλο των τοπικών φορέων. Έχει, είναι κάτι το πολύ σημαντικό και όταν είμαστε στον Ήγερα το έθιξαν αυτό. Που ξέφρασαν ε, λύπη από το του για όσα είχαν ε, συμφωνηθεί με τη Λιβύη ότι δεν εφαρμόστηκαν όπως πρέπει. Συμμερίζω με την αποψή σας ότι σε τοπικό επίπεδο επαρχίας εκεί αυτό θα πρέπει να προσέξουμε και να μπορέσουν να συμμετάσχουν οι πληθυσμοί οι ντόπιοι και να μην έχουμε έτσι μια μεθόδευση σε κεντρικό επίπεδο και μόνο. Και στις τρεις επισκέψεις μας σε αυτό επιμείναμε και να συναντηθούμε με τους νομάρχες, υπονομάρχες, αντινομάρχες κλπ. αλλά και με τοπικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών. Μακρά συζήτηση και, ε, που συνεχίζεται πάντα με τον κόσμο που συναντήσαμε εκεί και βλέπουμε ιδιαίτερη ζωντάνια θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε. Και στο σχέδιο αναπτυξής μας πολλά θα πρέπει να γίνουν ώστε αυτές οι τοπικές δραστηριότητες να ενισχυθούν. Το είπατε και καλά ότι ο Νίγηρας έχει μια μεταβατική κυβέρνηση που ανέβαλε και τις ε, εκλογές νομίζω και είναι υπεύθυνη πολιτική αποφασισμένη αλλά είναι αυτό το πούμε έτσι μια κυβέρνηση τεχνοκρατών που λέει εντάξει και οι επόμενοι την ίδια πολιτική θα ασκήσουν. Θα πρέπει να προσέξουμε ή από τώρα να προσπαθήσουμε με τους υπεύθυνους των πολιτικών κομμάτων η κυβέρνηση που θα βγει από τις δημοκρατικές εκλογές να ασκήσει την ίδια πολιτική. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για το θέμα της δημοκρατίας και την πολιτική της ε, Αλγερίας. Αντιμέτωπησαν ε, τρομερά πράγματα ε, εθνική σε εισαγωγικά καταστροφή έτσι γι' αυτό το να κάνω εγώ ένα σχόλιο τώρα δεν είναι και τόσο απλό αλλά αυτό που με εμπνέει είναι η προσπάθεια, προσοχή που αποδίδεται στα θύματα και στα Ηνωμένα Έθνη και στο ε, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε όλα αυτά και τα θύματα αυτά τότε υπάρχει πάντα παραμένει το πρόβλημα γιατί ε, για την εκπαίδευση των αστυνομικών αν είμαι υπέρ τώρα να έχουμε μια, μια προσέγγιση όχι μόνο στρατιωτική αλλά και με επιτόπου προσπάθειες είναι από τις χώρες στον κόσμο όπως το Αφγανιστάν εκεί βέβαια δικαιολογείται μια βάση αλλά εμείς είχαμε σαν προσέγγιση από ευρωπαϊκή πλευράς και από ποινική δικαστικής πλευράς είναι καλύτερη, ο καλύτερος τρόπος για να αγγιηθεί κανείς της ελευθερίας της ατομικής. Ε, ναι, εντάξει, υπηρεσίες πληροφοριών και σε αστυνομία. Επενδύσαμε πολλά, αλλά όχι ε, δικαστικά. Αν δεν οργανωθεί αυτό, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορούν να ξεφύγουν πολύ και εντάξει, καλύτερη εκπαίδευση των δικαστικών να γίνεται σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και να γίνονται σε αυτά τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, αλλά βέβαια και των θυμάτων. Έτσι θα έχουμε μια εγκύμηση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα για τη διαδικασία αυτή για την ρόλο των γυναικών να βοηθηθούν, ναι, υπογράφω, συνυπογράφω 1000% είναι σημαντικότατο για μια μετριοπάθεια, για την εκπαίδευση και όλα αυτά. Λοιπόν, για την εκπαίδευση και πάλι, αλλά θα το επιβεβαιώσει και ο συνάδελφος, η Ευρωπαϊκή Ένωση το προσέχει αυτό το θέμα ιδιαίτερα. Η κατάρτιση αστυνομικών και δικαστικών ε, να έχει και μια ιδιαίτερη πτυχή για την ε, σεβασμό και την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κι εγώ μερικά πραγματάκια. Για την τοπική αυτοδίκηση, τους τοπικούς φορείς πόσο συμμετέχουν, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του το είπε και ο κύριος Κερκόβε. Εδώ υπάρχει ένα κενό, το διαπιστώσαμε το κοινό. Και μας το είπαν οι ίδιες οι τοπικές κοινότητες οι επικεφαλής οι σοφοί, οι οποίοι μας μίλησαν για ενδογενείς λύσεις. Αυτό τον όρο χρησιμοποίησαν. Μας είπαν γιατί δεν μας βοηθάτε να εφαρμόσουμε δικές μας λύσεις. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει διαπραγματεύσεις. Στον Νίγηρα το πρόβλημα των εγκληματικών ενεργειών που επαναλαμβάνονται εμποδίζει τις προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Και είναι οι ίδιοι νέοι τους που είναι υπεύθυνοι. Οπότε αυτό το οποίο ζητούν οι τοπικές κοινότητες, οι κοινωνικές ομάδες, είναι να τις βοηθήσουμε να ξανασυνδεθούν με τους νέους, ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Είναι το κλειδί Οι σχέσεις επίσης των του ΑΡΕΚ με το κράτος στο Μαλί περνάνε μέσα από τις εθνικές αρχές, τις οικογενειακές αρχές, τις παραδοσιακές, που δυστυχώς βρίσκονται στο περιθώριο. Στο Μαλί και στον να το διαπιστώσαμε αυτό. Για την Αλγερία εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η Αλγερία. Συγχρόνως έχει και ένα παρελθόν που την κάνει να είναι δύσκολη η συμμετοχή της. Σίγουρα μπορεί θετικά να παρέμβει στο Σαχέλ, πολύ θετικά, μερικές φορές λιγότερο. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερο φως και περισσότερος διάλογος με τις διάφορες χώρες. Η ατιμορρησία, σίγουρα, πώς να βρει κανείς την καλή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη της συμφιλίωσης και την τιμωρία. Δεν πρέπει να υπάρχει ατιμορρησία. Εύκολα ερχόμαστε απ' έξω και λέμε «Α, πρέπει να γίνει αυτό ή να γίνει το άλλο. Πού είναι όμως τα όρια ανάμεσα στην τιμωρία και την ατιμορρησία. Η κάθε χώρα είναι καλύτερα σε θέση να βρει αυτά τα όρια. Εμείς πάντως δεν χρηματοδοτούμε την κατάρτιση στρατιωτικών. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ανθρώπους οι οποίοι να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για τη διάσταση της διακυβέρνησης, δίνοντας προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ισορροπία ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Θέλουμε στην αστυνομία να προσλαμβάνονται και οι γυναίκες, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για να βελτιωθεί η σχέση των δυνάμεων ασφαλείας με τον τόπιο πληθυσμό. Το βλέπουμε αυτό. Άρα χρειάζεται ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπωσδήποτε. Η Κομισιόν θέλει να χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα. Λίγα σχόλια για την περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία και την Αφρικανική Ένωση από τη σκοπιά των Ενωμένων Εθνών, όπως είπα, καταβάλουμε προσπάθεια να συνεργαστούμε με όλους τους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς παράγοντες, για παράδειγμα με την Αφρικανική Ένωση, για παράδειγμα με την ECOWAS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης εμπλέκεται πολύ στενά στην συνεργασία επίσης με το ε, Κέντρο Αφρικανικό Κέντρο που είναι εγκατεστημένο στην Αλγερία. Είναι ένας τρόπος λοιπόν ε, που προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις ικανότητες της Αφρικανικής Ένωσης και σε συνεργασία με την Αλγερία ο κλάδος μου προωθεί ένα ε, ε, σύστημα συνεργασίας τώρα. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε επίσης, όπως είπε ο Κέρκχοφ προηγουμένως, είναι ότι υπάρχει μια σημαντική χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Αφρικανικής Ένωσης, μια άλλη σημαντική χώρα η οποία δεν είναι μέλος της ΕΚΟΓΑΣ. Ο, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών βέβαια είναι ο οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν όλες αυτές οι χώρες και γι' αυτό ε, είναι, αυτός είναι μάλλον και ένας λόγος ε, για τον οποίο καλείται ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών να παίξει εκεί ένα σημαντικό ρόλο και να προσφέρει μια πλατφόρμα συνεργασίας. Αυτό που είδαμε και το βρίσκουμε και πολύ αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυση της συνεργασίας, ε, έχοντας δοσμένες τις δυσκολίες, είναι να αρχίσουμε από τα μικρά πράγματα. Μίλησα για την πλατφόρμα για την δικανική συνεργασία με συμμετοχή τεσσάρων κυβερνήσεων που ξεκίνησε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Αυτό απέρευσε από μια συνεργασία που είχαμε με μια χώρα. Όταν η χώρα αυτή εντόπισε ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει τη συνεργασία της, την δικανική συνεργασία δηλαδή με τις γειτονικές της χώρες και αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε με τρεις-τέσσερις χώρες στην περιφέρεια αυτή, στην περιοχή αυτή και αρχίζουμε σιγά σιγά να αναπτύσσουμε ικανότητα, capacity, η οποία ωφελεί επίσης και την συνεργασία και με άλλους εξωτερικούς φορείς. Επίσης, για την εκπαίδευση δεν εκπαιδεύουμε αξιωματούχους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ε, του αγώνα κατά της ε, εγκληματικότητας, αλλά αυτούς περισσότερο που είναι οι, ε, αυτοί που δίνουν τις οδηγίες για το πώς θα γίνει ο αγώνας αυτός, δηλαδή είναι πιο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Περί αυτού πρόκειται. Η προσέγγιση μας αυτή είναι και θεωρητική, αλλά και η εκπαίδευση δικαστών και εισαγγελέων ε, με αφορμή συγκεκριμένες υποθέσεις κλπ. Ο κλάδος πρόληψης τρομοκρατίας φτιάχνει τώρα ένα διδακτικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς με 10 διαφορετικά modules και αυτό για να καθοδηγούμε τους εκπαιδευτές οι οποίοι με τη σειρά τους θα προσφέρουν εκπαίδευση σε ε, εθνικούς φορείς. Και ε, το σύστημα αυτό θα μπορεί να προσαρμόζεται αναλόγως με τον φορέα. Ένα από τα μόντιουλ αυτά, ένα από τα τμήματα αυτά του προγράμματος αυτού θα έχει σχέση και με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με τα ανθρώπινα δικαιώματα που βεβαίως θα μπουν και ως mainstreaming σε ολόκληρο αυτό το ε, διδακτικό πρόγραμμα. Συγγνώμη, ένα ερώτημα. Είπατε ότι δεν εκπαιδεύει στρατιωτικούς με τα χρήματα της Επιτροπή. Δεν θέλω να κάνω στρατιωτικό κήρυγμα εδώ. Αλλά εκεί τα τρομοκρατικά, οι ομάδες, οι εγκληματικές ε, που είναι επιτόπου και πιο προχωρημένα μέσα έχουν, κυρίως μεταφόρας και χώρες αυτές Μαλή, ε, Νίγηρας, Μαυριτανία και περισσότερο δείχνουν ότι δεν έχουν δυνατότητες στρατιωτικές τους δυνάμεις για να ακολουθήσουν αυτούς τους τρομοκράτες ή εγκληματίες δεν έχουν το κατάλληλο υλικό, το κατάλληλο εξοπλισμό. Τι γίνεται και σε πτυχή συνεργασία, τι γίνεται. Δεν λαμβάνεται υπόψη λοιπόν αυτές, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτός ο στρατικός εξοπλισμός. Αυτή η συνεργασία είναι με χώρες σε διμερή σχέση όπως τη Γαλλία κλπ. Όχι στα πλαίσια λοιπόν μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Μήπως ε, θα μπορούσε κάπως να ελαφρυνθεί αυτός ο μηχανισμός για στρατικό μηχανισμό που δεν πάει για να σκοτώσει κόσμο όπως τα τζιπ ε, οχήματα παντός εδάφους, το ένα το άλλο και σε περίπτωση του και πώς θα μπορούσε κανείς να συνεργαστεί ολοκληρωμένα, προχωρημένα παρά με άλλες στρατηγικές σε διμερή βάση. Τι μπορεί να γίνει. Αν κατάλαβα καλά, αυτό το instrumental stability, αυτό το νέο ε, μέσο και εργαλείο θα χρηματοδοτήσει και αυτόν τον εξοπλισμό. Ε, καλά το κατάλαβα. Νομίζω ότι, εντάξει, ήμουν πολύ απόλυτο όταν είπα ότι δεν εκπαιδεύουμε στρατιωτικού. Δεν χρηματοδοτούμε την στρατιωτική κατάρτιση. Πληρώνουμε σε μερικές περιπτώσει για την κατάρτιση στρατιωτικών για αποστολέ. peacekeeping, για την ειρήνη, στην Αφρικανική Ένωση για παράδειγμα βοηθάμε σε περιφερειακό επίπεδο για τέτοιες ε, δραστηριότητες ή σχολές στρατιωτικών. Έμεσα δηλαδή χρηματοδοτούμε την κατάρτισή τους. Αλλά εννοείται ότι βλέπουμε τι περιλαμβάνει ακριβώς η κατάρτιση, έτσι ώστε να πρόκειται για την ε, προστασία της ειρήνης. Δεν χρηματοδοτούμε, εννοείται, να μάθει κάποιος πώς να χρησιμοποιεί ένα καλάσνικοφ ούτε και τον ε, εξοπλισμό ε, με όπλα των στρατιωτικών. Όχι. Έτσι κι αλλιώς, οι δαπάνες ελέγχονται και τα προβλήματα σε διεθνές επίπεδο δεν έχουν λυθεί ακόμα για το τι ακριβώς είναι συνεργασία στην ανάπτυξη όχι. Πάντως η Κομισιόν διαχειρίζεται μηχανισμούς στήριξης της ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ένδια και να έχουμε φόρα ανάπτυξη. Το θέμα της στάθμης και της ασφάλειας πάει πιο πέρα όμως και μας επιτρέπει δράσεις που ακριβώς μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της ασφάλειας. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα κάποιο πρόγραμμα όπου να χρηματοδοτήσαμε υλικό παρέμβαση εκτό μικροφώνου. Συνεχίζει ο κ. Λουί Μπλάνκο. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο στα πλαίσια τη σταθερότητα. Όχι. Αλλά μη σα πω και αν εσεί. Πρόεδρος, άλλος κανείς παρακαλώ. Παρακαλώ εσείς. Le recrutement de... Μιλήσατε για την πρόσληψη γυναικών στην αστυνομία. Πιστεύω ότι είναι εξαίρετη ιδέα. Όμως εδώ συμφωνώ με την κυρία Μπεναραμπάμ που αναφέρθηκε πριν στη σημασία που έχουν οι γυναίκες για την εκπαίδευση. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ καλό αυτό. Αναφερθήκατε επίσης και στο ριζασποστικό Ισλάμ στην περιοχή. Πώς όμως οι γυναίκες αυτές μπορεί να επιλεγούν για τέτοιες θέσεις ενώ ξέρουμε ποια είναι η θέση των γυναικών στο ριζοσπαστικό Ισλάμ που όπως είπατε και εσείς κερδίζει έδαφος. Ε, είναι πολύ δύσκολη η ερώτησή σας. Είναι αλήθεια ότι ο φανατισμός στο Ισλάμ οδηγεί στην μείωση ε, των γυναικών σε διάφορες σημαντικές θέσεις. Στην κοινωνία των Τουαρέκ όμως υπάρχει ο παραδοσιακός ρόλος των γυναικών όπου η γυναίκα έχει τη σκηνή. Αν χωρίσει από τον άντρα της, φεύγει με τη σκηνή της. Δεν ανήκει στον άντρα καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μια σημαντική δύναμη και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να διατηρηθεί αυτή η σχέση. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μόρφωση των γυναικών. Όπου υπάρχουν απειλές, όπως είναι στη Μαυριτανία, το στοιχείο αυτό κινδυνεύει. Για να καταπολεμήσουμε το φανατισμό στο Ισλάμ πρέπει να περάσουμε μέσα από την ενίσχυση των γυναικών στις παραδοσιακές κοινωνίες. Ωραία. Πρόεδρος, αυτά είναι και τα τελευταία λόγια στη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεισφέρατε στη συζήτηση ενός θέματος που προχωράει, που εξελίσσεται. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Θα σας ξαναχρειαστούμε θα παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση από κοντά. Να δούμε πώς η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, είπα εκπρόσωπος, που μπορεί να φροντίσει για αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνει και τι θα γίνει με, τις υπηρεσίες εξωτερικής, με την υπηρεσία αυτή, την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Δράση, όταν θα έχει ολοκληρωθεί, τι θα κάνει. Θα ανταλλάξουμε και πάλι απόψεις μεταξύ μας, ελπίζω, θα έχουμε την ευκαιρία και ελπίζω να ακούσουμε και την κυρία Άστον να έχουμε και από αυτήν στοιχεία για μια πραγματική ολοκληρωμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην περιοχή του Σαχέλ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα διακόψουμε για δύο λεπτά και μετά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Που έχει να κάνει με την ασφάλεια από τα χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο λεπτά διακοπή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 Ε, αυτά λοιπόν. Ε, να αρχίσουμε και πάλι. Να ξαναρχίσουμε και να τελειώσουμε για σήμερα. Να πούμε διάφορα πράγματα για το σχέδιο γνωμοδότησης που η κυρία Λέζιν ε, προετοίμασε σχέδιο γνωμοδότησης για την έκθεση της Επιτροπής αρμόδιας για την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδιο δρόσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Άννα Γκόμες, ε, είμαι στην Επιτροπή Ευασιών Ελευθεριών ε, εισηγήτρια. Κυρία Λέζιν, συντάκτρια οικονομοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα, επιθυμώ να σας Υποβάλλω το σχέδιο γνωμοδότησης για την χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα σας πω λίγο γιατί έγινε στο Shadow Meeting την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Πρώτα θα ήθελα να ε, αναπτύξω ε, τις εξής σκέψεις. Δηλαδή, πρώτα, η έκθεση της ΛΥΜΠΕ δεν είναι στη διάθεσή μας. Άρα, και για τη γνωμοδότηση, αλλά και για την παρούσα συζήτηση, στην πρώτη αυτή παρουσίαση στην ΣΕΝΤΕ, δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό το σχέδιο της ΛΥΜΠΕ, εφόσον δεν το έχουμε. Η πολιτική μου ομάδα και εγώ προσωπικώς θεωρούμε ότι χρειάζεται πάντοτε να διατηρείται μια αναλογικότητα ανάμεσα στην πραγματική απειλή και στα λαμβανόμενα μέτρα. Δεύτερο, ρίχνω ιδιαίτερο βάρος στην μη διάδοση, κυρίως ό,τι αφορά την υπογραφή και κύρωση των διαφόρων σχετικών συμφωνιών, εκεί όπου σημειώνονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι σε σχέση με την χιβιταροπή. Το τελευταίο μέρος της νομοδότησης περιλαμβάνει μια αξίωση της πολιτικής μου ομάδος, δηλαδή την σαφή διάκριση μεταξύ στρατιωτικής και μη στρατιωτικής χρήσης και για την αντιμετώπιση καταστροφών που θα πρέπει να έχει αποκλειστικά μη στρατιωτικό χαρακτήρα. Στην ε, shadow meeting που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πολλοί συνάδελφοι τάχθηκαν υπέρ τη συνεργασία μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού τομέα, πολιτική προστασία δηλαδή. Θεωρούμε εμεί ότι εάν επιτέλου η πολιτική προστασία εξοπλιστεί και από άψη προσωπικού και υλικού με τον τρόπο που απαιτείται, τότε θα μπορεί η αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών να γίνεται μόνο από την πολιτική προστασία χωρίς συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κίνδυνο που προέρχεται από βιολογικά όπλα, αναφέρομαι στην πράσινη βίβλο του 2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο, στην οποία βίβλο, κατά τη γνώμη μου, γίνονται πολύ ορθές προτάσεις. Για παράδειγμα, η ενισχυμένη εκπαίδευση του προσωπικού της πολιτικής προστασίας και το ξεκίνημα μιας διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών έτσι ώστε η πολιτική προστασία να είναι σε θέση να αναγνωρίζει όπλα βιολογικού χαρακτήρα και να γνωρίζει πώς πρέπει να αντιδράσει. Επικοδομητικές ήταν οι προτάσεις της ομάδας των Πρασίνων στην ε, διάρκεια της ε, σύσκεψής μας στο Στρασβούργο. Πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα στη γνωμοδότησή μου. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο του Παλέτσκης από τους σοσιαλδημοκράτες, με αυτό επίσης μπορώ να συμφωνήσω. Επίσης θεωρώ ότι τα όσα θίγει εκεί, εν μέρη τουλάχιστον περιλαμβάνονται στην γνωμοδότησή μου. Για παράδειγμα, ο, επαρκή, ο επαρκής εξοπλισμός της πολιτικής προστασίας. Ό,τι αφορά την κριτική τώρα σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα, σε ό,τι αφορά μια απογραφή την οποία ζητεί ο κ. Παλέτσκης για τα μέτρα που, είναι, που έχει στη διαθεσή της η πολιτική προστασία και στα όσα απαιτούνται, εγώ υπενθυμίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει περιεχόμενο γνωμοδότηση τη ΣΕΝΤΕ, την οποία συζητούμε τώρα. Και επίσης υποθέτω ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα περιλάβει ορισμένα σχετικά πράγματα στην έκθεσή της. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να παραπέμψω απευθείας στην έκθεση ΛΥΜΠΕ, αλλά όπως σας είπα δυστυχώς το κείμενο αυτό μου είναι ακόμη άγνωστο. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι για τις 16 Οκτωβρίου. Εφόσον έχουμε, ακόμα, εφόσον έχουμε μέχρι τότε μάλλον την έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Μου είπαν οι συντονιστές της ότι μάλλον θα υπάρχει μέχρι τότε. Εάν προκύψει ότι οι συνάδελφοί μας δεν προτείνουν ιδιαίτερα μέτρα για την ΧΒ τότε εγώ είμαι διατεθειμένη να συζητήσω εδώ με τους συναδέλφους μας, στην παρούσα επιτροπή δηλαδή, σχετικά μέτρα και να κάνω τις προτάσεις. Ευχαριστούμε. Η Άννα Γκόμες, ως εισηγήτρια από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά και εκ μέρου των σοσιαλιστών, μια που δεν είναι εδώ ο κύριος Παλέσκη. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Η κυρία Λούιζιν έχει δίκιο. Είναι παράδοξο Είμαι εισηγήτρια για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όμως σήμερα ολοκλήρωσα την έκθεσή μου, σήμερα την έδωσα στη μετάφραση. Κοίταξα το χρονοδιάγραμμα της ΛΥΜΠΕ και γι' αυτό δούλεψα έτσι. Αλλά βέβαια, στο μεταξύ, είδα γνωμοδοτήσει της κυρίας Λούζιν για παράδειγμα, το στο καλύτερο βέβαια και άλλων επιτροπών και τη Ήτρε. Και οι γνωμοδοτήσεις αυτές με βοήθησαν όπω καταλαβαίνετε να ολοκληρώσω το κείμενό μου, γιατί έτσι μπόρεσα να χρησιμοποιήσω κάποιε από τις ιδέες τους. Κάνοντας τη δουλειά αυτή για την ΛΥΜΠΕ, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέχασα ότι είμαι και μέλο αυτή εδώ τη υποπιτροπή. Προσπάθησα λοιπόν να ετοιμάσω μία πλήρη έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη και τις πτυχές της ασφάλειας και τις πτυχές της ελευθερίας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σύγκρινα. Γιατί βλέπετε, υπάρχει κάτι που ήδη από το 2009 έχει εγκρίνει τέλη του 2009 το Συμβούλιο. Σύγκρινα λοιπόν το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τότε με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι είδα? Ότι το Συμβούλιο αποδυναμώνει τις προτάσεις της Κομισιόν και μειώνει τις ευθύνες και των κρατών μελών και όλων σχετικά με το τι θα έπρεπε να κάνουμε ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κινδύνους από επιθέσεις τόσο βιολογικές όσο και ραδιολογικές, πυρηνικές και χημικές. Και το πιο σοβαρό είναι ότι στο μεταξύ, επειδή έχουμε τη Λισαβόνα, άλεξαν οι ευθύνε και αρμοδιότητες, γιατί έχουμε τώρα μια ρήτρα αλληλεγγύης. Είναι ευκαιρία λοιπόν αυτή τη ρήτρα αλληλεγγύης να την χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι και το νόημα της έκθεσής μου. Ζητάει από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το επίπεδο οριζόντιου συντονισμού που χρειάζεται ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, το οριζόντιο και το κάθετο, ανάμεσα στα διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. τίθεται θέμα ταχύτητας, αποτελεσματικότητας δράσης, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι. Δεύτερον, πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται η ανάλυση. Στη συνέχεια να γίνεται από κοινού σχεδιασμός, οι ε, δράσεις, επιχειρήσεις να σχεδιάζονται από κοινού. Και μετά μιλάω και για τους σπόρους. Έπειτα υπάρχει και το θέμα των συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει στη συνέχεια να ληφθούν ιατρικά κλπ. Ένα βασικό ζήτημα εδώ είναι να δώσουμε και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή υπάρχει στην πρόταση Επιτροπής, έναν κανονιστικό ρόλο και ρυθμιστικό ρόλο πιο σημαντικό από ό,τι έχει μέχρι τώρα. Και αυτό για να καλύψουμε τα διάφορα κενά οργάνωσης που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών. Σύμφωνο απόλυτα με την άποψη της κυρίας Λούζινγκ. Μιλάει για ενίσχυση των καθεστώτων μη διάδοσης. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Αλλά πρέπει να πάμε και πιο πέρα. Και γι' αυτό αυτός ο οριζόντιος και κάθετος συντονισμός είναι απαραίτητος. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε όλα τα προτινόμενα μέτρα. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, κάπου υπάρχει μια διαφορά με την προσέγγιση της κυρίας Λέζιν, η οποία βέβαια έχει διαφορετική οπτική γωνία. Όταν η κυρία Λέζιν μιλάει για πλήρη διάκριση της στρατιωτικής και της μη στρατιωτικής πτυχής, εγώ λέω ότι αυτό που χρειάζεται, το εδώ πέρα πρόκειται για τις ζωές των πολιτών. Πρόκειται για τις κοινωνίες μας, για τις υποδομές μας. Επειδή λοιπόν όλα αυτά διακυδεύονται, πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε διάρθρωση ανάμεσα στο στρατιωτικό και μη στρατιωτικό τομέα, είτε για την ανάλυση, είτε για τις πληροφορίες, είτε για την αντιμετώπιση. Είναι κεφαλαιόδου σημασία ο ρόλος ε, μηχανισμών. Αλλά για να είμαστε αποτελεσματικοί, και αυτό το ζητάω και το ζητάει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς παράγοντες που δεν αναφέρεται όπως πρέπει στο πρόγραμμα δράσης. Αυτή η διάρθρωση πρέπει να υπάρχει και με όλα τα κέντρα αριστείας, όπου τα κράτη-μέλη, όπως λέει και η κυρία Λιώσινγκ, είναι υποχρεωμένα να την έχουν για να καταπολεμηθούν βιολογικά χημικά όπλα. Αλλά η πραγματικότητα που ισχύει στα κράτη-μέλη για τον βαθμό με τον οποίο τηρούν τις υποχρώσεις τους στην πράξη, ο βαθμός αυτός διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πολλές χώρες δεν κάνουν αυτό που είναι υποχρεωμένα να κάνουν. Θα δείτε τις προτάσεις. Τέλη Σεπτεμβρίου έχουμε προβλέψει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την πρώτη συζήτηση. Βέβαια το κείμενο θα είναι έτοιμο νωρίτερα, θα το έχετε όλοι στη διάθεσή σας. Το Δεκέμβριο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλη, οπότε έχουμε καιρό για να ξαναδούμε όλες τις απόψεις και της κυρίας Λέζιν. Ο συνάδελφος Παλέσκης ο οποίος είναι υπεύθυνο από την ομάδα μου για να παρακολουθήσει την γνωμοδότηση της κυρίας Λέζινγκ μεταξύ άλλων, μου ζήτησε, επειδή δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, να τονίσω ότι οι επιθέσεις αυτές ή κυβερνοχώρο, για παράδειγμα, μπορεί να μην ε, έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες, αλλά η καταστροφή που θα προκαλέσουν είναι τεράστια. Γι' αυτό και πρέπει να γίνεται εξολόγηση κινδύνου κάθε τόσο. Επίσης, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για κινδύνους που έρχονται από κράτη, αλλά και εκτός κρατών, όπως μιλήσαμε πριν για την έρμο του Σαχέλ. Μου ζήτησε επίσης να σας πω και το εξής ότι χρειάζεται να αξιολογήσουμε και σε τι βαθμό είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απειλές από ιατρικής απόψεως. Επίσης, να δούμε τι δυνατότητες έχει η ενημέρωσης η Κομισιόν προς το Κοινοβούλιο. Πρέπει να γίνεται αυτή η ενημέρωση. Το λέω και εγώ στην έκθεσή μου. Γιατί στο κάτω-κάτω απορρέει από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, από το πρόγραμμα της Στοκόλμης κλπ. Χρειάζεται μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καλύπτονται τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο συμμετοχής των κρατών μελών. Επίσης χρειάζονται επαρκείς πόροι για να υπάρχει καλή προστασία των πολιτών και τέλος μιλάει και για την έννοια την εξής. Δεν πρόκειται μόνο για τη δράση μας άμα υπάρξει κάποιο συμβάν, ένα τύχημα ή μια επίθεση τρομοκρατική με χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά όπλα. Χρειάζεται να παρεύουν και στρατιωτικά τμήματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν με τη δικιά τους πραγματογνωμοσύνη. Τονίζει λοιπόν αυτή την ανάγκη καλού συντονισμού ανάμεσα στις γνώσεις που έχουν και οι στρατιωτικοί με τις γνώσεις που έχουν εμεί στρατιωτικοί. Ναι, από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκόμες μας διαβεβαίωσε ότι θα έχουμε το κείμενο στην Επιτροπή μας. Οπότε εντάξει. Για την Λέζιν, ε, το είπε η ίδια. Μίλησε για τον αφοπλισμό, την ε, διάδοση κλπ. και Πολλά και ωραία, αλλά δεν ταιριάζουν εδώ. Τα προβλήματα στην ανακοίνωση της Επιτροπής ε, όπως τίθενται δεν αντιμετωπίζονται. Αντίθετα, ε, και όπως λέει, με αυτό που είπε η κυρία Γκόμες, ε, το ξεπερνάμε ακόμα. Θέλω κάτι πιο ρεαλιστικό και οι τροπολογίες μου θα έχει να κάνει με όλες αυτές τις απειλές από το ξεκίνημα να δούμε πώς γίνεται, πώς μεταφέρονται, πώς αυτοποιείται το προσωπικό. Όλα αυτά τα πράγματα, όλη η αλυσίδα θα πρέπει να εξεταστεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με την κύριο Λεζίν, ε, για την πολιτική προστασία έχει ρόλο πραγματικά να παίξει περίπτωση καταστροφής. Ε, αν θέλουμε να πτύξουμε κάτι, καλό θα ήταν ε, βέβαια διαφοροποίηση από τον κύριο Λέζιν που αποκλεί οποιαδήποτε για πολιτικούς λόγους, μια οποιαδήποτε συνεργασία ανάμεσα στην πολίτες και στρατιωτικούς. Μήπως θα μπορούσαμε να δώσουμε το ένα μέσο για να αντιμετωπίσουμε παρόμοιο πρόβλημα. Θα πρέπει να συντονίσουμε τις δυνατότητες της προσφοράς απάντησης. Είναι σημαντικό κατά την απόψή μου. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τον πληθυσμό σε περιπτώσεις καταστροφής ή και να μπορέσουμε να δράσουμε τάχιστα, το είπε και η Χρειάζονται οι στρατιωτικοί, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, δεν είναι οι άνδρες, είναι η πείρα τους, η αναλύσή τους, το ένα το άλλο και χρειάζεται να συντονιστούν όλοι αυτοί για να βοηθήσουν τον πληθυσμό σε περίπτωση παρομοιου ατυχήματος, είτε με δόλο είτε όχι. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Και τώρα, εσείς. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία να αντιμετώπισε μια ιδιαίτερη κατάσταση τη στιγμή που χρειάστηκε να συντάξει την γνώμη της, ενώ η έκθεση δεν ήταν ακόμα στη διάθεσή μας τότε την ευχαριστώ για την προσπάθειά της, όπως επίσης και τα όσα προφορικά μας είπε μόλις η συνάδελφος Αναγκόμες. Ευχαριστώ και εκείνη. Έχει δίκιο ο κύριε Λόζεν που επιμένει ότι θα πρέπει οι προσπάθειες να συνεχιστούν για τη μια διασπορά παρομοίων όπλων ε, και όχι μόνο μία στον κίνδυνων, αλλά να εξαφανιστούν εντελώς τα πυρηνικά όπλα. Πάνω σε αυτό όμως η ομάδα μου δεν έχει ομόφωνη άποψη. Αν είστε όλοι υπέρ της μείωσης του ελέγχου, εντάξει, η ομάδα μου επίσης είναι υπέρ μιας αποπυρηνικοποίησης. Ε, δεν ξέρω αν είναι αυτό κάτι το ακρίβες, αλλά χρειάζονται για τον αφοπλισμό προσπάθειες να καταβληθούν με περισσότερο δυναμικό τρόπο, περισσότερο δραστήρια από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. όπως και άλλοι διαφωνώ με την ε, κυρία Λέζιν, γιατί επιμένει να ξεχωρίσει εντελώς τις στρατιωτικές ε, από τις δραστηριότητες των πολιτών ε, σε περίπτωση παρέμβασης, επανόρθωσης, εάν συμβεί κάτι, κάποια καταστροφή από όπου και να μας έλθει. Ήδη αυτά τα συζητήσαμε. Τα συζητήσαμε στην προπαρασκευαστική συνάντηση και σίγουρα ίσως έχει έτσι η κατάσταση που να απαιτείται μια στρατιωτική παρουσία ώστε να υπάρχει να εξασφαλιστεί έτσι μια ελάχιστη ασφάλεια ε, λόγω της παρουσίας της και μετά να προχωρήσουμε και στην επανόρθωση. Σίγουρα αυτό. Και όπως το είπατε κύριε μου, άδικο θα είχαμε να μην έχουμε υλικό και κόσμο με πύρα, ακριβώς στρατιωτικούς μας διαθέτουν πύρα και η χώρα μου έχει μια ειδική μονάδα την ε, ε τάχης της παρέμβασης που είναι εξειδικευμένη σε παρόμοιες ε, ε, επαναλαμβάνουμε παρεμβάσεις και σε ανθρωπιστικά θέματα και ε, δεν θα ήταν σωστό να μην τους χρησιμοποιήσουμε και τι έγινε ε, μήπως και εκτός από το Βέλγιο και η υπόλοιπη Ευρώπη θα έπρεπε να είχε μια παρόμοια μονάδα. Αυτό να ριωτιόμαστε σαν Βέλγοι. Πάντως ε, περιμένουμε ανυπόμονα το κείμενο που ε, μας υπόσχεστε κυρία Γκόμες για να μπορέσουμε να συντάξουμε τις ε, τροπολογίες μας από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Λέει ο κύριος μετά από τις πολύ λεπτομερείς δηλώσεις της κυρίας ε, Γκόμες αναμένω με ανυπομονησία την έκθεσή της σε ό,τι αφορά την έκθεση της Κελέσινγκ την έχω ήδη αναγνώσει και δεν έχω πολλά σχόλια να κάνω. Όπως είπε η κυρία Λέσινγκ, εμείς έχουμε υποβάλει ορισμένες συμπληρωματικές τροπολογίες, κυρίως εκεί όπου τίθεται το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας. Έχουμε ωστόσο και ορισμένες τροπολογίες δικές μας που θεωρούμε, όπου θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να δοθεί κάπως διαφορετικά το βάρος από ό,τι κάνει η κυρία για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το επίπεδο του κινδύνου όπου νομίζω ότι οι διατυπώσεις της κυρίας Λέζινγκ ενδέχεται να οδηγήσουν σε παρανοήσεις και ίσως είναι καλύτερα εκεί να τροποποιηθούν. Δεύτερο, όπου πρόκειται για θέματα απόσυρσης τακτικών πυρηνικών όπλων, νομίζουμε, η ομάδα των Πρασίνων και εγώ, Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να εμείνουμε, να εμείνουμε και στην απόσυρση πυρηνικών όπλων από το έδαφος της Δυτικής Ρωσίας, παραλίγο να πω ε, Σοβιετικής Ένωσης, αλλά κάπου η Ρωσία πάει να ξαναγίνει Σοβιετική Ένωση. Έχουμε λοιπόν και το αμφισβητούμενο, την αμφισβητούμενη παράγραφο 9 στην έκθεση της Λέζινγκ, όπου νομίζω ότι ενδεχομένως μπορούμε να συμβιβαστούμε. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει για κάθε νοητή περίπτωση να προβούμε σε χωρισμό και να απαιτήσουμε χωρισμό της στατιωτική από την πολιτική προστασία. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί σαφώς προτεραιότητα στην πολιτική προστασία, δηλαδή μη στατιωτική, και όχι να παραστήσουμε ότι δήθεν είναι αδιάφορο αν δράση θα αναλάβει η πολιτική προστασία ή κάποιο στρατιωτικό τμήμα. Αλλά νομίζω πάντω, όπω είπα, ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τι διατυπώσει ώστε να είναι αποδεκτέ από περισσότερου. Έχουμε... Άλλο κανεί που θέλει το λόγο. Να δώσουμε το λόγο πάλι στους συζητητές. Ε, η κυρία Λέζινγκ πρώτα απ' όλα. Ναι, πρώτα να καταστήσω σαφές ότι ο χωρισμός μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής προστασίας αποτελεί μια δική μας στόχευση. Είναι σαφές ότι εάν πρόκειται για μια ε, περίπτωση που μπορεί να συμβεί τώρα και όπου η πολιτική προστασία δεν διαθέτει πληροφορίες για την σύνθεση ας πούμε των βιολογικών όπλων, ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει κάποια συνεργασία. Ξαναλέω ότι πρόκειται για μια στόχευση δική μας, που σημαίνει βεβαίως ότι υπάρχει η προϋπόθεση ότι στο μέλλον η πολιτική προστασία θα πρέπει να εξοπλιστεί με τις ικανότητες αυτές. Σε ό,τι αφορά την διάδοση ή αν θέλετε τον εξοπλισμό και αφοπλισμό, επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι από τη δική μας σκοπιά απαιτείται απόσυρση όλων των πυρηνικών όπλων που θα σημάνει και μείωση του επίπεδου του κινδύνου, για παράδειγμα, από ενδεχόμενες τρομοκρατικές πράξεις που έχουν ε, στόχο πυρηνικά όπλα ή την χρήση τους. Άρα χρειάζεται ρίζοσπαστικός αφοπλισμός. Η κυρία χρειαζεται παστικος αφοπλισμος η κυρια γκομε ειπε και το επίπεδο πιθανότητας, ότι δηλαδή και ένα χαμηλό επίπεδο πιθανότητας μπορεί να έχει καταστροφικέ συνέπειες. Το γνωρίζουμε αυτό και είναι σαφέ. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε και στην αρχή ήδη του κειμένου μας ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ πρόκλησης, μεταξύ πρόκλησης απειλής και ε, αντίδρασης. Δηλαδή ανάμεσα στην επαγρύπνηση, ανάμεσα ενδεχομένως στο κράτος ή στις κρατικές δυνάμεις οι οποίες εποπτεύουν και μέχρι πού φτάνει αυτή η εποπτεία και στην αντίδραση. Τώρα μίλησε και για την ε, ρήτρα ελληνικής η κυρία Γκόμες. Και εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται συντονισμός των δράσεων ε, της πολιτικής προστασίας, εφόσον δηλαδή ε, χρειάζεται κάτι τέτοιο μεταξύ πολιτικών προστασιών πλειώνων χωρών. Επίσης από την πλευρά του Λαϊκού Κόμματος ακούστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λίστα. Εγώ όμως στις παραγράφους μου 5 και 6 ζητώ αυτή τη λίστα. Άρα δεν κατανοώ πολύ καλά το νόημα αυτής της ε, συμπληρωματικής παρατήρησης. Αυτά τα σχόλια έχω σημειώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, ναι, κάτι ξέχασα ακόμη. Για τη Ρωσία, ναι, είναι αυτονόητη η αξίωση αυτή, τα έχουμε συζητήσει ήδη στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ και συγγνώμη Δεν καταλαβαίνω την όλη διαδικασία στη συζήτησή με. Σαν σκιώδη συζητήτρια έλαβα αυτή την έκθεση, ξεκίνησα την ανάγνωση και είδα ε, για αυτά τα χημικά, βιολογικά κλπ. κλπ. και θα έπρεπε να δούμε τη σχέση και με το οργανωμένο έγκλημα, τι μπορούσαμε να κάνουμε, ένα ξεκίνημα επεξεργασίας απόψεων γι' αυτό. Αλλά χρειάζεται και χρειάζεται να περιμένω, χρειάστηκε να περιμένω την έκθεση και σήμερα το μεσημέρι που έφτασα την πήρα αυτή την έκθεση και δεν μπόρεσα να την αναγνώσω και στο ΕΛΚ δεν επεξεργαστήκαμε ακόμα το ποια θα είναι η στάση μας και δεν συζητήσαμε <laughs> νομίζω το συζητήσαμε για αυτά χημικά, βιολογικά, ακτινολογικά, πυρηνικά κλπ. Και αυτό δεν καταλαβαίνει τη σχετική διαδικασία. Εάν έχουμε μόνο μια εβδομάδα μπροστά μας για τις τροπολογίες, δεν επαρκεί. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς θα έχουμε το χρονοδιάγραμμά μας, πώς θα οργανωθούμε δηλαδή. Εδώ, παρόντες, συζητάμε, αλλά δεν διαβάσαμε την έκθεση. Την άποψη Τη ομάδα μου δεν τη γνωρίζουμε. Οπότε, καλύτερα να περιμένουμε. Εγώ δεν ξέρω για το ΕΛΚ, μη με ρωτάτε. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει άλλοι σκιώδες εισηγητές και πώς. Έτσι καλώ εξαρτόμαστε και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, γιατί η γνωμοδότησή μας θα ψηφιστεί εκεί. Οπότε ο καθένα έχει προθεσμίες που είναι σύντομε. Μίκαελ Γκάλερ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την σύντομη δήλωση της κύρια Γκόμες έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και πολύ στενά μάλιστα και για αυτή την συνεργασία μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού τομέα εμείς για λόγους συστηματικούς θα την υποστηρίξουμε. Εάν υποθέσω ότι μπορεί να υποστούμε επίθεση από κάποια τρομοκρατική ομάδα, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και το σχετικό υλικό είναι στα χέρια των στρατιωτικών δυνάμεων, είναι στα χέρια του στρατού. Αναγκαστικά θα πρέπει και η πολιτική προστασία να προσφύγει στη συνδρομή του στρατού. Ε, και εσείς το δεχθήκατε αυτό έμεσα. θα χαιρόμουν αν γράφατε στην πρώτη σας παράγραφο ότι για το λόγο αυτό, λέει στα αγγλικά, υποστηρίζει όλα τα κατάλληλα μέτρα, appropriate measures. Νομίζω ότι θα ήταν κατάλληλο, θα ήταν ορθή αυτή η διατύπωση και όχι μόνο civil measures. Ακριβώς επειδή τα πράγματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονάχα με τα μέσα της πολιτικής προστασίας. Ασφαλώς υπάρχει συμφωνία σε ό,τι αφορά την συμπλήρωση και ολοκλήρωση των διεθνών συνθήκων. Ε, όσοι δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει θα πρέπει να υπογράψουν. Αλλά σε ό,τι αφορά την αξίωση ταχύτητα του αφοπλισμού στην Ευρώπη, διερωτώ με γιατί άραγε η δημοκρατικότερη και πολιτικά σταθερότερη περιοχή του κόσμου να αφοπλιστεί εν ώψη ε, ενδεχομένων απειλών. Μα διότι μπορούμε, διότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή, λέει ο κ. Μπιουτικόφερ. Μα εγώ δεν το πιστεύω, απαντά ο κ. Γκάλερ, διότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν αυταρχικά καθεστώτα τα οποία θα παρανοήσουν την ενέργειά μας αυτή και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Εδώ πρόκειται για έκθεση επί μιας ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει θέσει το θέμα της αποπυρηνικοποίησης. Εγώ θα προτείνω η παράγραφος αυτή να διαγραφεί. Εάν βεβαίως δεν τα καταφέρουμε σε συμφωνία μαζί σας, τότε θα φροντίσουμε να υπάρξουν απαραίτητες πλειοψηφίες. Μια Μιας και εγώ έγραψα το κείμενο στα αγγλικά, μπορώ να το δώσω ευθύ αμέσω ε, στους συναδέλφους που ε, θα ήθελαν να το διαβάσουν στα αγγλικά. Ε, άλλωστε τα αγγλικά μου θα χρειαστούν κάποιες διορθώσεις από τους μεταφραστές και θα πρέπει να μεταφραστεί και όλα στο κείμενο. Ήθελα να πω ότι βεβαίω μπορεί να συζητηθεί το θέμα Πρόκειται για έκθεση για λογαριασμό της ΛΥΜΠΕ. Δεν συζητώ λοιπόν θέματα τοποθεσίας πυρηνικών όπλων. βεβαίω και είμαι υπέρ του αφοπλισμού, αλλά δεν ε, είναι θέμα της παρούσης εκθέσεως. Μιλούμε για το σχέδιο δράσεως, δηλαδή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι είναι διατεθειμένη και έτοιμη να πράξει σε περίπτωση μιας τρομοκρατικής επιθέσεως και όχι μόνο για επίθεση με πυρηνικά όπλα, αλλά και ραδιολογικά, βιοχημικά κλπ. Εγώ ζητώ την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντίδρασης σε κρίσεις με συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών μέσων για την καταπολέμηση, για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε καταστροφής αροβιταχή ατομικών, ραδιολογικών, βιοχημικών όπλων. Έχουμε ωστόσο ένα μηχανισμό που είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή έχουμε πει τα σχετικά και στο ψήφισμα ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να, να, να μπορεί να φροντίσει να δοθεί άμεση συμπαράσταση, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα αλλά και εκτός εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η χρήση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, των υφιστάμενων δομών δηλαδή, θα πρέπει η χρήση αυτού του μηχανισμού να γίνεται για μια ανταπόκριση σε τέτοια πρόκληση. Αλλά υπάρχει και το προηγούμενο στάδιο του εντοπισμού των κινδύνων και της ε, προπαρασκευής. Εκεί χρειάζεται συνεργασία και με τις στατιωτικές ε, δυνατότητες. Διότι ένα μέρος των operators είναι μη στατιωτικοί. Είναι για παράδειγμα ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή ραδιοβιολογικών ή πυρηνικών υλικών τα οποία ενδεχομένως μπορεί να κλαπούν από κάποιους ε, εγκληματίες. Και ε, βεβαίως αυτοί εμπλέκονται και σε θέματα μεταφορών τέτοιων υλικών κλπ. Είναι λοιπόν κρίσιμο το θέμα αυτό το οποίο ήδη θίγεται στο σχέδιο δράσεως και θα πρέπει να ενισχυθεί. Α, λοιπόν, να λοιπόν ένα ακόμη στοιχείο το οποίο προτίθεμαι να περιλάβω. Βεβαίως η συζήτηση μόλις τώρα αρχίζει. Οι συνάδελφοι όπως η κυρία Λέζινγκ, αλλά και άλλοι που έχουν απόψεις θα τις παρουσιάσουν στη διάρκεια ε, των συζητήσεων και στην παρουσία Επιτροπή αλλά και στην Επιτροπή ε, Θεμελιωδών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών να πάει στις 28 Σεπτεμβρίου και έτσι να έχετε μπροστά σας στη διάθεσή σας δύο εβδομάδες να επανεξετάσετε το σχεδογνωμοδότηση, να συντονιστείτε στις ομάδες σας και την τρίτη λοιπόν το μεσημέρι έτσι τα από την Ολομέλεια του Στρασβούργου και έτσι να παρακολουθήσετε την κατάσταση και να συντονιστείτε, να οργανωθείτε έτσι, έτσι και να προετοιμαστείτε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. επανέρχομαι στα επιχειρήματα ορισμένων συναδέλφων που είπαν ότι τα όσα διαλαμβάνονται στην παράγραφο 4 του σχεδίου εκθέσεως της κυρίας Λουέσινγκ, δηλαδή το θέμα της απόσυρσης πυρηνικών όπλων, δεν θα έπρεπε να ενταχθεί στο παρόν σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ένα κείμενο γενικότερου χαρακτήρα για τέτοια θέματα που να μην περιλαμβάνει και την αξίωση απόσυρσης των πυρηνικών όπλων. Θα θυμίσω τον κάτω να τον πρεσβύτερο που έλεγε πάντοτε, όχι κάρτακο τελέντα έστα, αλλά τα πυρηνικά όπλα πρέπει να καταστραφούν, παραφράζει ο κ. Μπιτικόφερ. Εντάξει, σε αυτή τη γλώσσα και η τελική φράση, έτσι, τελευταία λέξη. Αρκούμεθα σε αυτά σήμερα. Κάτι για την οργάνωσή μας. Επόμενη συνάντηση 27 Σεπτεμβρίου. Κρίστιαν Χέλλερ που συνεργασία στρατητικό πολιτική. Έτσι πριν από τις καλοκαίρι το είχαμε εξετάσει αρκετά. Θα πρέπει να δούμε και πάλι τι θα γίνει με την προθεσμία της τροπολογίας. 28 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τρίτη, με την ΕΦΕΤ έχουμε τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, σημαντική συνάντηση, γι' αυτό σας παρακαλώ παρόντες και να λάβετε και το λόγο για να υποστηρίξετε τις θέσεις μας, οι οποίες 28 ναι, οι οποίες ε, κινδυνεύουν να στριμωχτούν άσκημα από τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτά. Η Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ Έχουμε από εκεί μια παρέμβαση από την Γραμματεία του ΝΑΤΟ στη συνάντησή μας με, τους, ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Γεια σας.